Dear colleagues, ladies Αγαπητοί συνάδελφοι. Η ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Διότι έχουμε εδώ την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το οποίο αποτελεί τον, το σημείο υπαρχμών 6 της ε, εμείς για την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις δικαστικές υποθέσεις. Με χαρά μας σας ξαναυποδεχόμαστε κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Ρέντιν, για αυτήν ε, την ευκαιρία που θα έχουμε τώρα μαζί σας να δούμε τα θέματα της ε, σχετικής πολιτικής. Αλλά, βέβαια, έχουν προκύψει και ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες κάποια σημαντικά. Είμαι βέβαιος ότι είστε σε ετοιμότητα για, την, ε, για τις επαφές αυτές με Ηνωμένε Πολιτείε. Μια από τι τελευταίες εβδομάδες, με μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθήσαμε τα σχετικά με το PRISM. Αυτό το πρόγραμμα ασφαλείας που αφορά την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, που φυσικά ε, συνεπάγεται σημαντικά για τις σχέσεις μας και κυρίω για την ε, συνάντηση της 13ης ε, Ιουνίου μεταξύ ημών και εκείνων σε επίπεδο Υπουργών Δικαιοσύνης. Θέλουμε επομένω και, και, και εγώ μας να τα συζητήσουμε αυτά μαζί σας. Και περιμένουν πώς και πώς κάποιοι συνάδελφοι εδώ. Μια που ανοίγουν στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Και ενώ τον συνάδελφο Έλερ. Κύριε Επίτροπε, θα σας δώσουμε το λόγο και κατόπιν θα ακολουθήσει η συζήτηση. Πάντως ε, είμαι βέβαιος ότι κυρία Αντιπρόεδρε γνωρίζετε πόσο μας έχει προβληματίσει αυτή η υπόθεση. Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Και οι πολίτες αυτοί με τα λόγου γνώσεως προβληματίζονται και θέλουν πληροφορίες. Τι γίνεται με, τις, ε, με τον ιδιωτικό τους βίο και ζητούν οι αρμόδιες αρχές να τους προστατεύσουν. Έχετε τη σκητάλη κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα εδώ για αυτήν την τακτή ανταλλαγή απόψεων, τον διάρθρωμενο διάλογο που και έτσι μπορούμε να κάνουμε ε, αυτή την επισκόπηση όλων των ζητημάτων που μας ενδιαφέρουν Νομίζω και χέρι-χέρι πετύχαμε πάρα πολλά και πρόκειται τώρα για το χρονικό περιθώριο το οποίο έχουμε, τόσο ώστε να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία έχουμε αναλάβει. Να σας ε, πω επίσης ότι έχουμε αυτή την οδηγία την οποία και θα καλείστε να ψηφίσετε. Ε, η κυρία Αντωνέσκου είναι η συγκήτριά σας και θα την συγχαρώ για το έργο που επετέλεσε, διότι σε συνεργασία με τους χιόλους εισηγητάς ε, κατέληξε σε αυτό το πάρα πολύ φιλοδοξό κείμενο, μια που αφορά αυτά τα δικονομικά δικαιώματα, τόσο σημαντικά για τους Ευρωπαίους. Όπως σας έχω υποσχεθεί, θα συνεχίσω το έργο μου όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα, την νομική αρρωγή, τους ε, ευάλωτους, τους, τους μη προνομιούχους τέλο πάντων υπόπτους σε σχέση με το τεκμήριο της αθωότητος και το ότι έχουμε επιτελεί σημαντικό έργο δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα να σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε. Επίσης δε, όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε με το, το πακέτο τη δέσμη μέτρων που αφορούν τα μέτρα για το, τα θύματα, τους παθόντες έχει νομοθετήσει το Συμβούλιο κατόπιν των δικών σας προτάσεων και τώρα έχουμε περάσει στη φάση της ε, υλοποίησης της εφαρμογής. Όμως έχουμε επιτελέσει και έργο στο πεδίο του ποινικού δικαίου για να προστατεύσουμε τις κοινέ αξίες, τα αγαθά, ούτω ώστε κάποια σοβαρά εγκλήματα θα εντοπίζονται, θα ορίζονται στην ποινική τους υπόσταση και θα διώκονται μιλήσαμε για την παραγάριξη του ευρώ, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, πρόκειται για τα χρήματα των φορολογούμενων, τα οποία καταλήγουν στις λάθος τσέπες, τσέπες των εγκληματιών. Έχουμε μπαίνει σε αυτό το νομοθέτημα του Κοινοβουλίου, ε, αυτό γίνεται στα πλαίσια της πολιτικής για την προστασία των οικονομικών συμφωνών της Ένωσης, σε επίπεδο ε, ποινικού δικαίου. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει το καθήκον του, όπως ε, πάντοτε το πράτεται, και ότι έτσι θα υλοποιήσετε τις αρχικές μας φιλοδοξίες και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτόν τον δημιουργικό διάλογο μαζί σας και με το Συμβούλιο Οπότε έχουμε αυτό το νομοθέτημα. Αυτό θα το ε, αναλάβει η Λιθανική Προεδρία που θα πάρει τη σκητάλη και πριν από τα τέλη του έτους ελπίζουμε να έχουμε κλείσει αυτό το κύκλο και ε, αυτό το τονίζω διότι η αδίποτε καθυστέρηση ωφελεί τους εγκληματίες. Έχουμε επίσης και τα θέματα του Ευρωπαίου Ισαγγελέως για τις ε, έρευνες, την ποινική δίωξη όσον αφορά τα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφωνών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας παραβέβω στο άρθρο 86 της Συνθήκης. Ο Ισαγγελέας θα στέλνει την προσοχή του στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και επίση θα δούμε κατά πόσο δυνατόν να έχουμε μια ολοκληρωμένη, σφαιρική αλλά και αποκεντρωμένη ε, αντιμετώπιση, ένα σύστημα ολόκληρο σε σχέση με τα όσα θα αναθέτει ο Ευρωπαίο Αγγελέα στους Εθνικού Αγγελείς. Αυτά όσον αφορά ε, κάποιες ε, ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά την ανεξαρτησία, όσον αφορά ε, ε, να μην υπάρχει εξάρτηση από θεσμικά όργανα και από εθνικές αρχές. Και έτσι να υπάρχει αξιοπιστία, έτσι να υπάρχει νομιμοποίηση και παράλληλα βέβαια να είναι υπόλογος της οπότε θα πρέπει και το Κοινοβούλιο τελικά να αξιολογήσει τις επιδόσεις, θα πρέπει να διέπεται από δικαστικό έλεγχο και επίση να υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ δικονομικέ εγγύσει. Όλοι αυτοί οι κανόνε είναι ξεκάθαροι και επίσης όπως ισχύουν και αλλού θα πρέπει να ισχύουν και για τον Ευρωεισαγγελέα. Επίση θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου μη γραφειοκρατική δομή σε αυτή την υπηρεσία όπω το προβλέπει η συνθήκη και έτσι θα πρέπει να μπορεί να γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση. Επομένω, θα πρέπει να έχουμε γραφειοκρατικό άθο ε, Οπότε τελικά θα πρέπει να μπορεί να επικεντρωθεί αυτή η υπηρεσία ει το βασικό καθήκον της. Η Eurojust βεβαίω και είναι μια αξιόλογη υπηρεσία, αλλά θα πρέπει επίσης να λειτουργεί πιο εύρεθμα. Τώρα, όσον αφορά την ε, πολιτική για τα ναρκωτικά, έχουμε παρουσιάσει κάποιε νομοθετικέ προτάσει και έχουμε τώρα μια, ένα νέο νομοθέτημα για τι ψυχοενεργητικέ ψυχοενεργητικές ουσίες και έτσι να μπορέσουμε ε, να έχουμε μια πολιτική πιο βιώσιμη Η επί. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και όσον αφορά την καταπολέμηση των δυσμενοδιακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τον ε, ε, φροντίζει για την ένταξη στην κοινωνική των Ρωμά και θέλουμε τώρα τα κράτη-μέλη επίσης να υλοποιήσουν, να προχωρήσουν τις εθνικές στρατηγικές στα πλαίσια της δικής μας ε, πολιτικής. Επίσης υπάρχει μια πρόταση σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά την ε, κοινωνική ένταξη των Ρωμά. εκεί είναι οι εξή. Πρώτα-πρώτα πρόσβαση στην ε, παιδεία, την απασχόληση, την υγεία και τη στέγαση. Και επίση να έχουμε κάποιο είδου ε, εγκάρσια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, όπω ε, η κατάσταση των ανηλίκων, των γυναικών, η διασυνορική συνεργασία και ο γενικό στόχο είναι να έχουμε πιο αποτελεσματικό έργο ή στα κράτη-μέλη. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, η οποία αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρώμα, θα λάβει μέρο στο συμπόσιο στι 27 έκτο, οπότε πρόκειται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μα του ανηλίκου και του νέου. Και θα δούμε τι θα γίνει με τι κοινότητε των Ρωμά και θα συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη. Η κυρία Γιαρόκα πρόκειται να αντιπροσωπεύσει το Κοινοβούλιο στο συμπόσιο αυτό. Όπω ακριβώ ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε τι αιτήσει εκθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την υλοποίηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, σας δείχνω εδώ την έκθεση για το 2012. Εκεί καλύπτουμε τις εξελίξεις κατά το, το, το έτος. Επίσης έχουμε μια συστηματική η υλοποίηση αυτού του χάρτη. Όμως για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει δουλειά πολιτική, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος πολιτικός και νομικός, τόσο ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις εφαρμογής των δικαιωμάτων. Η φετινή έκθεση δε ε, στέκεται και τονίζει την υλοποίηση του χάρτη αυτών των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε τα δικαστήρια να παραπέμπουν και να ζητούν μια προδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως βλέπουμε ότι έτσι προσφεύγουν τελικά ή στον χάρτη και αυτό παναδεί ότι όλο ένα και περισσότερο ριζώνει στο μυαλό των εθνικών δικαστών η ύπαρξη αυτού του χάρτη. Και είμαι θα και κοινότητες δικαίου, επομένως. Δεν μπορούμε παρά να βασιζόμαστε, να πρέπει να βασιζόμαστε στα εθνικά δικαστήρια. Οπότε οι εθνικοί δικαστές ε, μπορούν να εγγυηθούν το ότι θα απολάβουν τον δικαιωμάτων τους οι Ευρωπαίοι. Επομένως, συμβάλλουν στο να έχει κάποια συνέπεια το σύστημα αυτό και έτσι να έχουμε την προστασία των δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα κοινοτικού δικαίου. Τον δε Μάρτιο, όπω γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, ξεκίνησε αυτή την, την καταγραφή των επιδόσεων. Τον πίνακα βαθμολόγιο όπω το λέμε όσον αφορά τα θέματα της δικαιοσύνη που είναι ένα εργαλείο το οποίο ε, εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το καταρτήσαμε αυτό, τόσο ώστε να έχουμε αξιόπιστα, συγκρίσιμα, αντικειμενικά δεδομένα για την λειτουργία των ε, συστημάτων της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη. Και στις 29 Μαΐου, όπως ξέρετε, ε, έχουμε κάποιες ε, συστάσεις που διατυπώσαμε συγκεκριμένα σε κάθε κράτο μέλος. Και έτσι είπαμε θα πρέπει να κάποια μέτρα ώστε να βελτιωθεί η οικονομία της δικαιοσύνης. Γενικά το δικά σύστημα σε κάθε χώρα μέλη και έτσι να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο για μας είναι μια προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα για αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οπότε και όλοι θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι πρόκειται για κάτι το οποίο το ζητούσαν έκαθεν το Κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί. Ξέρω ότι εγκρίνατε την έκθεση Ταβάρες και προσπαθήσατε να δείτε πώς το κράτος δικαίου θα διαφυλαχθεί καλύτερα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως αυτό είναι ζήτημα πάρα πολύ βασικό και γι' αυτό και είναι σημαντικό όλα τα δεσμικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη να εμπλακούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο επ' αυτού. Ας θυμηθούμε την ομιλία Μπαρός που πέρσι είχε ζητήσει καλύτερα μέσα πολιτικής, σε καλή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίστηκε, δούλεψε πάνω σε αυτό και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης στις 6 ε, ψήφισε κάποια συμπέρασματα και είπαμε ότι το 2013 θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή οπότε θα πρέπει να δούμε και το ότι τα συμπεράσματα, τα βάρες αποτελούν μια ουσιαστική συμβολή σε αυτή τη διαδικασία που θέλουμε να φέρουμε εις πέρας. Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας έχουμε οργανώσει τέλος Αυγούστου ένα σχετικό σεμινάριο και επίσης θεωρούμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε αυτή τη διάσκεψη για τη δικαιοσύνη ε, όπου θα συμμετάσχουν ε, δικαστές, διάφοροι εμπλεκόμενοι, πολιτικοί, για να συζητηθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ο Πρόεδρός σας έχει βεβαίως προσκληθεί. Επίσης, Θεωρούμε ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται στις προσδοκίες των πολιτών. Βεβαίω, οι πολίτε προσδοκούν και την προστασία των δεδομένων του. Γιατί, όταν μιλούμε για θεμελιώδη δικαιώματα, μία από τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι και η προστασία αυτών των προσωπικών δεδομένων. Άρα, το κοινοβούλιο τώρα επιτελεί ίσως το σημαντικότερο από αυτής της με την έκθεση που επεξεργάζεται. Οπότε, όπως ξέρετε, σε σχέση με το πρίσμ <clears throat> έχει υπάρξει μεγάλος προβληματισμός και έτσι είδαμε ότι η προστασία των δεδομένων δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Αυτό κατέδειξε επίσης ότι μόνο με κάποιο, κάποιο στεγανό σύστημα προστασία μπορεί να αποδώσουν να διηγήσουν στην, στην εμπιστοσύνη των πολιτών που να πιστέψουν ότι είναι προστατευμένοι. Σε σχέση τώρα με τις ε, αποκαλύψεις των ΜΜΕ για το πρίσμ, στις 10 Ιουνίου υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων προς τους Αμερικανούς. Απίθυνα μια επιστολή στον Eric Holder που είναι ο Γενικός Αγγελέας. Ακόμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης βέβαια δεν μου έχει απαντήσει, αλλά τα είπαμε και στην Υπουργική Σύνοδο στο Δουβλίνο. Και εκεί διατύπωσα τις ε, επιφυλάξει μου σε σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών και ε, ζήτησα διευκρινήσεις. Επίσης, έθεσα το ζήτημα των διαφορετικών επιπέδων προστασία όσον αφορά αυτά τα ε, προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή το τι ισχύει από τη μία μεριά του Αμερικανού πολίτε και από την άλλη μεριά το τι ισχύει για του Ευρωπαίου πολίτε τη Ένωση αυτό το θέμα. Πανελειμμένα η φυγεί εδώ. Σε σύμπτωτη δίκαιο διέπει τις ε, εταιρείες που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολλές φορές είναι ασαφές το αν έχουν αρμοδιότητα για τις υποθέσεις τους τα Αμερικανικά ή τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Αυτά είπα στον εισαγγελέα Χόλτερ, ή στον υπουργό τέλο πάντων Χόλτερ. Ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε την κατάσταση έτσι, ώστε να μην ε, έχουμε την ε, διάπραξη κάποιων ε, ενεργειών, κάποιων, μην έχουμε κάποιες πράξεις οι οποίες συμβαίνουν στο κοινωτικό δίκαιο. Αποφάσισα λοιπόν να δημιουργήσουμε μια διατλαντική ομάδα με τον Eric Holder για να συζητήσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης ζήτησα ε, να γίνουν ενισχυμένε προσπάθειες για να φτάσουμε σε συμφωνία για την ομπρέλα προστασία των δεδομένων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΗΠΑ που θα εξασφαλίζει ε, ίδια προστασία για τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών με των Αμερικάνων πολιτών. Δεύτερον, τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να χαίρουν τις ίδια ελάχιστη προστασία με των Αμερικάνων πολιτών και πιστεύω ότι είναι και η ώρα να σημειώσουμε πρόοδο στη διαπραγματεύση στο θέμα αυτό. Και τώρα περνάω στην ε, δική μα γενική πρόταση για την προστασία των δεδομένων, που είναι σημαντικό τμήμα τη απάντηση και που θα βοηθήσει για να επιλύσουμε τι ε, νομικέ αβεβαιότητε για τι εταιρείε που συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες και επιλέγουν να συμβαστούν το δίκαιο της μίας του ενός μέρους, αλλά κινδυνεύουν να παραβιάσουν το δίκαιο του άλλου μέρους. Με τη νέα πρόταση ε, προωθούμε διάφορα μέτρα. Ε, ρητή συνένεση καταρχάς, είναι προϋπόθεση. Επίσης, τι γίνεται με τις αμερικανικές εταιρείες δραστηρίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Όταν, ακόμα και όταν τα προσωπικά δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι ήταν ένα καμπανάκι αυτό που έδειξε σε όλους, η πρόταση αυτή ήταν ένα καμπανάκι που έδειξε σε όλους πόσο επίγον είναι να προχωρήσουμε με ένα ισχυρό νομοθέτημα και στον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα της εφαρμογής του δικαίου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ωφελήσει ε, όλους εκείνους που δεν θέλουν να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων τους. Και τώρα, Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω τις δηλώσεις που έκαναν πολλοί ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες που ζήτησαν να επιταχυνθεί η διαδικασία. Θα ήθελα να σας πω, Πρόεδρε, ότι για αυτό το θέμα μας παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Αν θα κάνουμε κάτι, προσπαθεί να δει και πώς θα το κάνουμε. Γιατί αν καταφέρουμε αυτοί οι κανόνες προστασίας να συμφωνηθούν, τότε θα έχουμε δημιουργήσει ένα χρυσό κανόνα για την προστασία των δεδομένων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας μην χάσουμε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία. Ευχαριστούμε για τις δηλώσεις σας, για τις χειρές δεσμεύσεις σας, για τα τόσο σημαντικά θέματα που συζητάτε στο διάλογο με τις ΗΠΑ. Όπως είπατε, όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας, αλλά πιο πολύ είναι σημαντικό το βλέμμα των Ευρωπαίων πολιτών, που ανησυχούν για το τι γίνονται τα προσωπικά τους δεδομένα δεν εφαρμόζεται κανένας ε, κανόνας ό,τι αφορά την επεξεργασία τους. Ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται πέστε. Ούτε κανένα άλλο δίκαιο. Η συζήτηση λοιπόν έχει ξεκινήσει. Έχουμε ένα κατάλογο πολλών ομιλητών, 20 τουλάχιστον ομιλητέ. Έχουμε μια μισή ώρα για τη συζήτηση αυτή, όπως συνέβη και σήμερα το πρωί όταν ήταν παρόν ο Έλληνα υπουργό. Θα δώσω το λόγο σε τουλάχιστον 20 ευρωβουλευτέ. Σα σας παρακαλώ και κάνω έκκληση να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Ε, με ευελιξία μένα, αλλά δύο λεπτά δε. Και μετά να έχει το χρόνο και η Επίτροπος να απαντήσει. Ας ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, με την κυρία Ματιό που είναι συντονίστρια του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπη, σε ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα είμαι λακωνική, έχω τέσσερα σημεία να θέσω. Θα ξεκινήσουμε το ΠΡΙΣ. Αυτό που συμβαίνει είναι σοκαριστικό, πρέπει να το πω. Έχετε δίκιο, Επίτροπε, που υπενθυμίζετε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία και στον κανονισμό και στην οδηγία ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί κάτι δεν έκαναν καλά και πρέπει να το υπενθυμίσουμε εδώ. Καλό είναι που δημιουργήσατε μια ομάδα εργασίας διατλαντική με εμπειρογνώμονε. Εντάξει, καλό είναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο στενάροι από αυτό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να πέφτουν θύματα κατασκοπίας ε, και τα προσωπικά τους δεδομένα να φεύγουν προς ε, τις Πολιτείες. ακόμα και αν είναι θέμα εσωτερικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος Ομπάμα μας εξηγεί βέβαια ότι με αυτόν τον τρόπο ε, καταπολεμάει την τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο όπλων, αλλά εμείς στο βαθμό που δεν έχουν ακόμα συναυθεί οι συμφωνίες πρέπει να έχουμε στεναρή στάση και ακόμα δεν έχουν συναυθεί οι συμφωνίες. Όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων, αυτή η διατλαντική ομάδα, προχωρήσει τις εργασίες της. Ελπίζω, κυρία Επίτροπε, να μας εξηγήσετε πώς ε, προχωρούν αυτές οι εργασίες και τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Ένα άλλο ερώτημα που με απασχολεί τα μάλλα. Όπως και πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές μπαίνω στο Twitter και βλέπω ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν ρατσιστικά σχόλια, αντισημητικά και κατά των ομοφιλοφίλων ε, στο site hashtag. Πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να επαναφέρουμε στην τάξη αυτό το site, γιατί αυτά που λέει είναι όλο και πιο απαράδεκτα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έπειτα, και τελευταίο πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα ξέρετε ότι την Παρασκευή στη Σόφια Ο κύριο Πέσκι, ε, επικεφαλής των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών, θα είναι επικεφαλής μάλλον των μυστικών υπηρεσιών, άτομο που είναι λίγο αμφιλεγόμενο, μαφιόζος από ό,τι φαίνεται. Ε, πολλοί ε, έκαναν διαδηλώσεις στη Σόφια. Τι γνώμη έχετε. Και επίσης για τους Ρώμα και την ε, ένταξη των Ρώμα στη Γαλλία. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες ό,τι αφορά τη μοίρα των, Ρώμο, των Ρώμα. Είναι στις ειδήσει στη Λιόν, ας πούμε, είχαμε δύο θανάτους. Ένα κλειστό εργοστάσιο πήρε φωτιά, πυρκαγιά ήταν. Επίσης, ε, ρίξανε βόμβες Μολότοφ σε στρατόπεδα, σε καταβλισμούς Ρωμά. Τι σκοπεύετε να κάνετε εναντίον της ε, γαλλικής κυβέρνησης που δεν προστατεύει επαρκώς τους Ρώμα. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεδομένης και της χρονικής πίεσης, πολύ λυπάμαι που, που δεν μίλησε η κυρία Ρέντινγκ για όλα τα θέματα. Να σημειώσω ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για το Ρωμά, όπου και θα πρέπει να δείξουμε πώς αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη το θέμα των μειονοτήτων. Πρωτού ζητήσουμε το οτιδήποτε από τρίτα κράτη μέλη, από τρίτα κράτη. Να επικεντρωθώ στο θέμα όμως που έχει να κάνει με τις ε, θεωρήσεις, το οποίο και θέλουμε να συζητήσουμε. Κάποιοι είπαν ότι, κοιτάξτε, αυτά τα ξέραμε πάντα. Αυτά που εμένα με ενοχλούν και είμαι από το 2009 εδώ στο Κοινοβούλιο και από την αρχή μου λέγανε ότι οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, είναι σημαντικοί εταίροι μας και θα πρέπει να είναι η συνεργασία μας μια συνεργασία εμπιστοσύνης, αμοιβαίας. Του προσπάθησα λοιπόν αυτό. Αν όμως αυτοί οι φίλοι και οι εταίροι με τους οποίους συνεργάζομαι σε καθεστώς αμοιβαίου σεβασμού ε, μυστικά καταχράζονται, καταχράζονται τα δεδομένα των πολιτών μας χωρίς να μας ενημερώνουν, θεωρώ, ότι είναι δραματικό το ζήτημα. Και δεν στέκει ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την δίωξη ποινικών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας. Οι δημοσιεύσεις, σε σε διάφορα έντυπα μέσα καθιστούν σαφές ότι γενικά υπάρχει μία παρακολούθηση, ελέγχεται μετανάστευση και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Και έτσι έχω περάσει λοιπόν στο θέμα της προστασίας των δεδομένων. Αναρωτιέμαι αν όντω πρέπει να βιαστούμε σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία. Ερωτώ Μήπως οι συζητήσει θα πρέπει να περιλάβουν και διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία θα ασκήσουν κριτική στην πολιτική αυτή συμπεριφορά αλλά θα δημιουργήσουν και κανόνες προκειμένου τουλάχιστον να μην επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Να είναι σαφές ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα ισχύουν. Και ξέρω ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Ο Αμερικανός πρόεδρος ε, λέει ότι κοιτάξτε αγαπητοί πολίτες της Αμερικής δεν πρέπει να ανησυχείτε, αυτό αφορά μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε. Τι λέμε δηλαδή, ότι μη ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να μαζέψουμε δικά σας στοιχεία, θα μαζέψουμε δεδομένα άλλων πολιτών. Στη Γερμανία είχαμε και ένα σχέδιο κατά της δημοκρατίας. Καλό ήταν αυτό στη θεωρία αλλά συμπεριλάμβανε και πολίτες οι οποίες έμεναν τυχαία δίπλα σε κάποιον ύποπτο. Γι' αυτό λοιπόν είναι δραματικό αυτό το ζήτημα και κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Και τέλος, ένα τελευταίο σημείο, θα ήθελα να καλέσω την Επίτροπο να μείνουν από κοινού σε ό,τι αφορά την επεξεργασία τους η οδηγία και ο κανονισμός ότι πρόκειται για την προστασία των δεμένων των πολιτών μας σε κάθε κατάσταση της ζωής τους, ακόμα και αν υπάρχει υποψία από άλλα μέλη. Ευχαριστώ κυρία Ιντφέλτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την εισαγωγή της. Δύο θέματα θα ήθελα να δείξω. Το ένα ήταν το μου, ασφαλώς, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Όπως είπε η κυρία Σίπελ, ήμουν από εκείνους που εξ αρχής ε, έθετε επανειλημμένα, πραγματικά τόσα πολλά χρόνια επανειλημμένα ε, ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής και συνεχώς μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα λυθούν όλα με τη νέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και κοιτάξτε πού καταλήξαμε. Σε μια κατάσταση σύμφωνο με αυτά που είπε η κυρία Σίπελο, οι ιδιαίτεροι φίλοι μας, αν θέλετε, και εταίροι μας, δεν μας αντιμετωπίζουν με φιλικό τρόπο, αλλά σαν υποπτούς. Και να ασκήσουμε κριτική στους Αμερικανούς, σύμφωνοι, αλλά να ασκήσουμε κριτική και στον εαυτό μας, γιατί οι Αμερικανοί μας, οι Αμερικανοί θα μας εκμεταλλευτούν όσο τους αφήσουμε. Και οποιοδήποτε άλλος δηλαδή. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει λίγο πιο πολύ χαρακτήρα και να πει στους φίλους και εταίρους και ιδιαίτερα σε χώρες που δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εταίροι ποια είναι τα όρια μας. Και δεν είναι και η πρώτη φορά, ξέρετε, το 2006 επίσης καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή η, ε, υπόκλεπταν τα δεδομένα SWIFT των τραπεζών επί σειρά ετών. Και τώρα δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ξεχάσουμε ε, το τι έγινε μετά από κάποιο καιρό και σε λίγα χρόνια θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση ή θα διευκρινίσουμε στους Αμερικάνους ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το άρθρο 42, το πρώην άρθρο 42 στο σχέδιο κανονισμού. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι θα επανέλθει στον κανονισμό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εξηγήσει γιατί μεταξύ του πρώτου σχεδίου το οποίο διέρευσε, όπου υπήρχε αυτή η ρήτρα, το άρθρο 42 και του επίσημου σχεδίου το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο ε, εξαφανίστηκε το άρθρο αυτό. Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί εκείνοι που διόρθωναν το κείμενο, ποιοι το διόρθωναν, γιατί αφαιρέθηκε αυτό, αυτή η ρήτρα και τι θα κάνουμε για να επανέλθει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι η Συμφωνία Safe Harbor ουσιαστικά έχει αφαιρεθεί, δεν έχει, έχει μείνει κενή και δεν λειτουργεί. Και τέλο τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Υπάρχει μια μεγάλη μειονότητα στο α, κοινοβούλιο που έχουν ζητήσει 11 φορέ διασφάλιση των δικαιωμάτων. Και σε ό,τι αφορά το σχέδιο ε, δράση τον οδικό χάρτη. Και στο Συμβούλιο πλέον το ζητούν αυτό πολλά κρατημέλη. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε, και για τα δικαιώματα πάλι των σεξουαλικών μειονοτήτων. Η επόμενη Προεδρία είναι της Λιθουανίας. Στα τέλη Ιουλίου θα γίνει το Gay Pride στο Βίλνιο, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Δεν έχει απαγορευτεί αυτή αυτό το Gay Pride, αλλά έχει εκδιωχθεί, αν θέλετε, έξω από το κέντρο της πόλης και αναφέρεται ότι δεν μπορεί να ε, βεβαιώσει, να διασφαλίσει η αστυνομία ότι μπορεί να προστατεύσει μια τέτοια διαδήλωση. Μα αν δεν μπορεί η αστυνομία να, δια, να προστατεύσει μια τέτοια ειρηνική διαδήλωση, πώς πρόκειται να προστατεύσει μια τέτοια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως να μην κάνουμε τη σύνοδο αυτές στο Βέλγιο, η κυρία Σαντζεντίνη. Um... I was still in... Ε, να, να πάρω το μικρόφωνο γιατί α, α, ήθελα να απολαύσω τις τελευταίες φράσεις της Σοφίνετ Φέλτ αλλά πάντως θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να, να, να, να, να αντιμετωπίσουμε ε, αυτό που είπατε, αυτό το χάρτη των επιδόσεων για την δικαιοσύνη και επίση να δούμε τι θα γίνει με το εμπορικό δίκαιο, τι θα γίνει με το διοικητικό δίκαιο, πώ θα τα συνδέσουμε για αυτά με αυτή την υπόθεση και βέβαια θα πρέπει η νομική επιτροπή μα να ασχοληθεί με αυτό. Αλλά όμω από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνα, δημοκρατία, κράτο δικαίου και όλα αυτά, η συνθήκη λέγοντα τα θεωρεί ζητήματα που είναι ε, συναρμοδιότητα της Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, σας ερωτώ κυρία Επίτροπε, πώς Σκοπεύεται να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή του ΣΥΠΗΝ ε, αυτού του, του, του, χάρτη επιδόσεων του Σκόρμπορ για να μπορείς να καλύψει το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα κλπ. Και επίσης να δούμε το πώς θα υπάρχει καταγραφή κράτος μέλος των όσων γίνονται. Και να καλύψουμε και τα ζητήματα εμπορικού δικαίου αλλά και διοικητικού δικαίου. Κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά αυτή την νομική αρρωγή, Τώρα αξιολογούμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, προγραμματίζουμε για το μέλλον. Αλλά η πράσινη θεωρούμε ότι η αδίποτε συνεργασία για ποινικό δίκαιο και δικαιοσύνη δεν είναι δυνατόν να θεωρείται κάτι ξεχωριστό από την νομική ρογή. Το άσυλο, το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψης, δεν υπάρχει δικαιοσύνη χωρί νομική αρρωγή. Επίση θα πρέπει να ξεκαθαριστεί που δεν έχει γίνει ακόμα το να υπάρχει μια ε, πραγματική ολοκληρωμένη πρόταση πάνω σε αυτό. Η σχετική συνεργασία δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν νομοθετήσουμε για την νομική αρρωγή. Μας αναφέρατε γιατί τι με τον Υπουργό Χόλτερ. Όσον αφορά το πρίσμα, όσον αφορά την προσέγγιση των δεδομένων. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πρόεδρε, κλείνω, κλείνω. Αναφέρατε ότι συναντήσατε κάποιου εμπειρογνώμονε, κάποιου ειδικού από Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τη ΣΥΠΑ, ώστε να ξεκαθαριστούν όσα εκκρεμούν. Ποιοι είναι αυτοί, είναι γνωστοί, μπορείτε να μα πείτε ποιοι είναι αυτοί οι επαείοντε του οποίου συναντήσατε. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κέρκο που έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για το πρίσμα, να πούμε δύο λόγια, γιατί ακούσαμε τις απόψεις άλλων συναδέλφων, ακούσαμε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι αρκεί εγώ να σας πω ότι γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν πληροφορίε και τεχνολογία κατά τον κόσμο οι εγκληματίε, οι οργανωμένοι αλλά και οι τρομοκρατέ. Επομένω, βεβαίω και είναι θεμητή προσδοκία το να χρησιμοποιείται η τεχνολογία κατά αυτόν. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σύνομο θα πρέπει να γίνεται με τον σεβασμό του δυτικού βίου και κυρίως εμείς να προσέξουμε το δυτικό βίο των Ευρωπαίων του οποίους και εκπροσωπούμε. Θα πρέπει να μπορούμε να συλλέγονται τα δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την Επιτροπή και την Επίτροπο που προσπαθούν επομένω κάτι να ε, διεξέλθουν, κάτι να διεκπαιρεώσουν και οπότε θα πρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω το εξή κυρία Ρέντι. Πρόσφατα, ορισμένοι εξημών πήγαμε αποστολή στην Σουηδία να εξετάσουμε κάτι το οποίο έχει σχέση με τους ασυνοδεύτους ανηλίκους. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία καταλήγουν στη χώρα εκείνη. Αλλά και σε άλλα κράτη της περιφερειάς τη Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω. Συχνά προέρχονται από τρίτε χώρες, οι γονεί του απλά τα εγκατέλειψαν αλφαβήτα λόγο και λέμε ότι ανέζητουν ένα καλύτερο αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό το κάνουν και για άλλους λόγους που δεν είναι και τόσο παραδεκτή, αποδεκτή. Και κάθε πρέπει να αξίζει γιατί τα φροντίζουν αυτά τα παιδιά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το ότι οι γονείς οι οποίοι απαρνούνται τις ευθύνες τους κάνουν κάτι το οποίο κατά τη γνώμη είναι ανήθικο. 100% απαράδεκτο. Οπότε παρακαλώ θέλω να ακούσω τη γνώμη της κυρίας Επιτρόπου. Τι πρεσβεύει. Πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ώστε να εξασφαλίζει ότι οι γονεί δεν θα απαρνούνται τις ε, ευθύνες τους με αυτόν τον απεχθή τρόπο. Κύριε Μπρόντσο. Όποτε έχουμε κάποια διαφορά, κάποια προστριβή μεταξύ δύο αντιδίκων και ε, θα πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια όσον αφορά το, το, το πώς θα ιεραρχηθούν αυτά τα αντιμαχόμενα δικαιώματα. Επίσης ανέφερε κύριε πίτροπος, το είναι σημαντικό να κατησχύει το, το, το, το, το κράτος δικαίου και να το σέβονται όλα, όλα τα θεσμικά όργανα. Συμφωνείτε επομένως ότι από την άλλη μεριά έχει το κάθε κράτος το δικό του δίκαιο, αλλά έχουμε και τυραννικά κράτη. Τι, τι γίνεται με αυτό. Και οπότε πολλές φορές έχουμε κάποια νομοθετήματα τα οποία βασίζονται σε κάποια ιδεολογήματα και ουσιαστικά καταρρύπτουν το κράτο δικαίου. Άρα και σπαραμένουμε στο άρθρο 21 του Χάρτη Δικαιωμάτων. Αν επομένω ε, έχουμε το άρθρο 21 το οποίο ορίζει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε δυσμενεί διακρίσει επί τη βάση των πολιτικών πεπιθήσεων. Τι θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά κάποια κράτη τα οποία απολύουν κόσμο ε, και κυρίω τον απολύουν από το δημόσιο, διότι ε, αυτοί οι απολυόμενοι ανήκουν σε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Τέλος, έχουμε κάποια νομοθετήματα σε πολλά κράτη που απαγορεύουν το φιλετικό μίσος, ε, απαγορεύουν την, ε, ε, την υπομόχλευση, τέλος, την υποδάβληση αυτού του, του, ρατσιστικού μίσους. Οπότε δεν θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και στο να μην έχουμε αναμόχλευση παθών επί τη βάση πολιτικών διαφορών. Και αυτό δεν το κάνουν ούτε οι πολιτικοί όμως. Και τώρα το λέω θα ο κύριος Έλλερ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής μας ε, της, της, της αντιπροσωπείας μας ε, για τις ΗΠΑ. Κύριε Έλερ, έχετε το λόγο. Θα Πρόεδρε, ότι έγινε αυτή μας η, η, η αποστολή, απευθύνθηκαμε σε εσά και ε, αντιδράσατε αμέσως, ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε επίσης τον τον, τον διατλαντικό, υπερατλαντικό διάλογο. Αλλά όσον αφορά αυτό το διάλογο έχουν νομική βάση οι Αμερικανοί. Και καταλαβαίνω ότι τώρα είναι συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα και ότι θέλετε κάτι να πετύχετε. Οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιδράσετε επί τη βάση ένστασης κατά αυτής της νομικής βάσης που έχουν οι Αμερικανοί. Και όσον αφορά τον διατλαντικό και ατλαντικό διάλογο, διαμορφώσαμε αντίστοιχα την ημερησία μας διάταξη. Θα βάλουμε και αυτό το θέμα επομένω, το πρίσμα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ενημέρωση μαζί σα. Οι Αμερικανοί λένε όμω από την άλλη μεριά ότι το πρίσμα είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Άρα να φροντίσουμε όχι μόνο να έχουμε πυρομαχικά εισαγωγικά για τι επαφέ με του Αμερικανού, αλλά ίσω θα πρέπει να προβληματιστούμε για το τι είναι εφικτό, τι είναι πρακτικό. Το φθινόπωρο θα ξανασυντηθούμε με τους Γερμανούς. Οπότε όλα αυτά πρέπει τότε να ληφθούν υπόψη. Και παρακαλώ και θέλαμε για τη δική σας βοήθεια, για τις πληροφορίες αυτές που μας είναι χρήσιμες. Κύριε Φώσου. Σας ευχαριστώ καταρχάς και εγώ έχω δύο σημεία τα οποία ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς το σε αντιμετωπίζουν και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταρχάς το είδαμε και το ακούσαμε παντού. Η κατάσταση στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αποδεκτή. Θεωρώ ότι υπάρχει και μία έλλειψη συμφωνιών. Και θα έλεγα επί της αρχής και ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μας ότι εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε και δύο αρχές. Καταρχάς, χωρίς πρόσβαση, χωρίς νομική βάση και κατά δεύτερον τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών ε, όταν τα επεξεργάζεται κανείς θα πρέπει να τηρεί και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Η λύση δεν μπορεί να είναι, θεωρώ, να μεταφερθεί το πρόβλημα στις εταιρείε. Θα πρέπει κυρίως να πετύχουμε μια συμφωνία για την προστασία των δεδομένων. Το αναφέρατε και θεωρώ ότι τα διεθνή πρότυπα και οι κανόνες για την μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να είναι κάτι το εφικτό. Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα, θεωρώ για το μέλλον, θα είναι να επιλύσουμε, να ρυθμίσουμε πού βρίσκονται τα σύνορα, τα όρια για την συλλογή ιδιωτικών στοιχείων. Ε, ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς προκειμένου να είναι αξιόπιστο το σύστημα της προστασίας των δεδομένων και προκειμένου να ε, εμπνέει η εμπιστοσύνη. Δεύτερη ερώτηση τώρα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για ένα σημαντικό φάκελο, ένα σημαντικό θέμα για την πιο στενή αστυνομική και δικαστική συνεργασία και θεωρώ ότι όλο και πιο πολύ μας οδηγεί σε θέματα αντιμετώπισης, εγκληματικότητας και σε σε αρμοδιότητας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Ρωτώ λοιπόν πότε θα δούμε την πρόταση αυτή. Πόσο, τι παιδί εφαρμογής θα έχει και ποιο ενδιαφέρον ίσως Πού θα έχει έντρα η Ευρωπαϊκή Δικαστική Εποπτεία. Με ποιος, με άλλα λόγια, ποιος θα αποφασίζει αν κάποιος θέλει να καταγγείλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή. Ευχαριστώ κυρία Ρωμέρα Λόπας. Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Είναι ευθύνη της κυρίας ε, Μάλτσρομ βέβαια αυτό. Όλοι οι πολίτες περιμένουν τα αποτελέσματα. Και είναι στον πυρήνα της διατλαντικής ατζέντα μας αυτό το θέμα. Ίσως έχουμε διαφορετικές στρατηγικές ε, εμείς και οι Αμερικανοί για το πώς καταπολεμούμε τον, την τρομοκρατία. Ε, και ίσως δεν τις γνωρίζουμε αυτές τις διαφορές. Ε, καταρχάς έχουμε διαφορετικές απόψεις για το πώς αντιμετωπίζουμε την ιδιωτική σφαίρα. Θεωρούμε ότι είναι φοβερή παραβίαση της ιδιωτικής μας σφαίρας μόνο και μόνο για λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ένας Ισπανός χιουμορίστας λέει ότι όταν ε, κατεβαίνουμε στους δρόμους ε, δεν μας ακούνε. Όταν καθόμαστε σπίτι μας κατασκοπεύουμε, μας κατασκοπεύουν. Αυτή την κατάσταση ζούμε δηλαδή. Αυτή την κατάσταση ζούμε εδώ στην Ευρώπη. Σαν να έχουν βγει οι μπάτσοι στους δρόμους και να μας κατασκοπεύουν. Τελικά η Ευρώπη τι σημαίνει. Δεν αισθανόμαστε προστατευμένοι, δεν αισθανόμαστε σωστά πλαισιωμένοι, αισθανόμαστε προδομένοι. Κυρία Ρέντιν, το βασικό είναι αν θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μας δώσει απάντηση. Πρέπει να ενημερωθούμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα ε, για ενημέρωση. να σταματήσουν αυτές οι ιστορίες με τους εμπειρογνώμονες. Όλο δημιουργούμε ομάδες εμπειρογνωμόνων και στο μεταξύ δεν μας δίδονται αποτελέσματα και απαντήσεις. Ευχαριστώ την ε, Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ που είναι παρούσα. Είμαι σχεδόν ηγήτρια των φιλελεύθερων για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Και φυσικά ε, πρέπει να θέσω διάφορα θέματα. Φυσικά θέλω υψηλά επίπεδα προστασία στον κανονισμό, αλλά φοβάμαι ότι η η μεγαλύτερη ιστορία είναι ότι η Κομισιόν στο σχέδιο ε, κειμένου της δεν έβαλε τη ρήτρα 42 που έλεγε ότι καμία απόφαση δικαστηρίου και καμία απόφαση δικαστικής αρχής, ε, διοικητικής αρχής δεν θα χρειάζεται για δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα εφαρμόζεται με κανένα τρόπο. Εσείς αυτή τη ρήτρα την ξεχάσατε ρίξατε βόμβα στις διαπραγματεύσεις. Θα δεχτείτε τώρα την επανεισαγωγή στον κανονισμό προστασίας των δεδομένων της ε, ρήτρας αυτής. Εγώ και η Σόφη Ιντβελτ θέτουμε ερωτήματα εδώ και χρόνια για αυτά τα ζητήματα. Έγινε μια συζήτηση πριν από 18 μήνες στην Ολομέλεια. Και τότε και σήμερα μας είπατε ότι πρέπει να πιέσουμε μέσω των συνήθων καναλιών, αλλά δεν χρησιμοποιούνται αυτά, δεν γίνονται σεβαστά. Το ξέρετε εσείς και το ξέρουμε και εμείς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς μας φέρατε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και τέλος πάντων, τώρα, τι προοπτικές υπάρχει για αυτή τη συμφωνία τη διατλαντική και θα θα καλύψει και τις εξουσίες για θέματα πληροφοριών. Αυτή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ που προστατεύει την, τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών από την ανάμειξη των υπηρεσιών πληροφοριών. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές ε, θα δημοσιοποιούνται, τα στοιχεία που μας δίνουν οι Αμερικανοί μπορούν να δημοποιηθούν. Ο κ. Ευχαριστώ για την προστασία ε, προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών θέλω να μιλήσω. Μετά από αυτές τις ιστορίες που αποκάλυψαν ε, την, ε, το πρόγραμμα παρακολούθησης της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, της NSA, Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των αρμοδιοτήτων και του ελέγχου σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα θεσπίσουμε κανόνες στην Ευρώπη για τις υπηρεσίες πληροφοριών ε, τις υπηρεσίες εδώ στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά δεν έχουμε αρμοδιότητες προς το παρόν. Αλλά θέλω να μιλήσω και για την ε, συμφωνία πλαίσιο, γιατί συνδέεται με αυτήν. Θέλω ως εισηγητής να ζητήσω τα θεμελιώδη δικαιώματα να υπάρχουν, να υπάρχει το δικαίωμα ένδικων μέσων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να το θέσουμε αυτό το θέμα άμεσα και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα τους κανόνες για τις υπηρεσίες πληροφοριών όσο δεν μπορούμε, τότε θα πρέπει να δώσουμε ε, τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να προστατεύουν τα δικά τους δεδομένα. Η αλλαγή στον κανονισμό που τόνισε η κυρία Λάτφορ, ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση αν ε, υπάρχει μεταφορά σε δεδομένων σε αρχές τρίτης χώρας, είναι πολύ σημαντική αυτή η αναγνώριση. Μην ξεχνάτε ότι το Yahoo, το Google κτλ. Ε, δίνει τεράστιους όγκους προσωπικών δεδομένων ε, από εδώ και από εκεί. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να ξέρουν ε, ή να δίνουν τη συγκατάθεσή τους στα δεδομένα που επιθυμούν να διαβιβαστούν κτλ. Μην ξεχνάμε το επίπεδο προστασίας της οδηγίας του 95. Τουλάχιστον αυτό το επίπεδο να κρατήσουμε. Είναι σημαντικό ελπίζω και προσβλέπω στην ε, υποστήριξη της Κομισιόν και για το Συμβούλιο θα να πω τα εξή. Από ό,τι ακούω από το Συμβούλιο, υπάρχει μια είναι λίγο ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστική κίνηση για τον κανονισμό και για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν υπάρχει κίνηση, δηλαδή, ενώ αλλαγή της τάσης του Συμβουλίου. Θα ήθελα να πιέσετε λοιπόν εσείς από πλευρά Κομισιόν το Συμβούλιο να αλλάξει στάση. Ο εισηγητή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τον καονισμό προστασίας των δεδομένων είναι ο επόμενος ομιλητή. Α, συγγνώμη, μίλησε. Ο κύριος Ντρούτσας θα μιλήσει τώρα για την οδηγία. Θα είμαι σύντομος γιατί οι συνάδελφοι με κάλυψαν στα περισσότερα. Και εγώ με τη σειρά μου εκφράζω την ανησυχία μου για αυτά που συμβαίνουν. Να χρησιμοποιήσω τα λόγια της κυρίας Ρέντινγκ στη δική της παρέμβαση. Δηλαδή ότι οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις για τις ΗΠΑ Πολιτείες είναι το καμπανάκι αφύπνισης για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες και όσου ασχολούνται με την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μάθημα που πρέπει να μάθουμε είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στην ε, μέχρι τη δυνατή προστασία των δεδομένων αυτών στην, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και δυνατόν να το αυξήσουμε αυτό το επίπεδο προστασία. Και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Γιατί εδώ μιλάμε για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και πώ θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Αυτό πρέπει να ακούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στη δική μου πολιτική ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, αυτό επιδιώκουμε. Ελπίζω ότι και άλλες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου θα κατευθύνονται, θα καθοδηγούνται από αυτές τις αρχές, να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις προσπάθειές της και ας πάω τώρα στην οδηγία. Την ευχαριστώ που επανεπιβεβαιώνει την στεναρή της θέση, επιμένει στην προσέγγιση του πακέτου γιατί τα μηνύματα που έρχονται από το Συμβούλιο, αλλά πρέπει να πω και από άλλες πολιτικές ομάδες δυστυχώς στο Κοινοβούλιο είναι ανησυχητικά. Δεν πρέπει να θυσιάσουμε την οδηγία μόνο και μόνο για να πετύχουμε, να έχουμε κάτι σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων. Ευχαριστώ. Ο, κ. κύριος ασχολείται επίσης με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, yes, ε, I... Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπέ Ρέντινγκ. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είμαι εισηγητή τη Επιτροπή Ήτρα για την προστασία, για τον κανονισμό για την προστασία και φυσικά μέλο τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Είπα. Από κάποιε απόψει θα ήταν καλή χρονική συγκυρία, ίσω ε, αυτή. Γιατί ξεκινάμε τι διαπραγματεύσει με του Αμερικανού για το TTIP για το πακέτο για τις επενδύσεις και για την εταιρική σχέση και δεν έχουμε επίση ολοκληρώσει την ε, νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων των πολιτών μας. Έχουμε λοιπόν ε, σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Σε ένα χρόνο τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά ίσως. Κατά δεύτερον, το βασικό ζήτημα θεωρώ είναι το εξή. Αυτό που είπε η Επιτροπή Ρέντινγκ, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ίση αντιμετώπιση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον είπα. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας. Θα πρέπει να το διασφαλίσουμε. Αν θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε το άρθρο 42, θεωρώ ότι αυτό θα έκανε πολλά για να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά θα υπάρχει συντιμετώπιση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσει η προτεραιότητά μας. Επίσης, να το τονίσω αυτό, θεωρώ το ανέφερε και ο κ. Κερχόπη και ένας άλλος συνάδελφος, ο λόγος που παρουσίασαν οι Αμερικανοί που, για, τον, για το ότι πέρασαν αν θέλετε τα νόμιμα όρια είναι η προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας η οποία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη γι' αυτό λοιπόν δεν είναι απλό να την καταπολεμάει κανείς είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει όμως με νομική βάση και αυτή αποτελ... αυτό αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση και για τις ε, αρχές του ε, ΗΠΑ και για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είμαστε μπροστά από τους τρομοκράτες, τηρώντας όμως παράλληλα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας και πάντα να τηρείται η νομίμη βάση. Λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία μέσω του TTIP και του κανονισμού να τα πετύχουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Sogor. Thank you. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Αμερικανοί φίλοι άλλαξαν το σλόγγαν, δεν λένε Yes we can, λένε Yes we can». Σαρώνουμε. Με όλον το σεβασμό προς την Επίτροπο θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι μόνο προσωπικό. Δεν θεωρείτε ότι στο μέλλον θα πρέπει να αναθεωρήσετε και να ζητήσετε να συμμετέχετε, να συμμετέχετε σε όλες τις μυστικές συναντήσεις όπως τελευταία στην Bilderberg και πρόσφατα, μάλλον σήμερα αναφέρθηκε η Daily Telegraph σε εσά και χτες ε, ο εκπρόσωπός σας ε, δεν απάντησε, δεν αρνήθηκε άμεσα τις κατηγορίες αυτές που σας ε, απευθυνθήκαν. Απαντήστε αν θέλετε. Δεν διαβάζω την Daily Telegraph, λέει η κυρία Ρέντινγκ, η Επιτροπή, Ρέντινγκ, τι ακριβώ ανέφερε. Εκτό μικροφώνου, ο κύριο Σίγκορ. Yes, yes. Ο κύριο Σόγκορ, ναι. Θέσετε το ερώτημά σα ξεκάθαρα, λέει ο πρόεδρο. Μιλήστε, ίσως, μιλάτε ίσως με τον εκπρόσωπό σας. Χτες ε, ένας ε, δημοσιογράφος της Daily Telegraph μετά από ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ρώτησε κατά πόσο αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι θα αναμειχθείτε στις εκλογές του επόμενου έτους στην Ουγγαρία και δεν αρνήθηκε την κατηγορία αυτή ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να σχολιάσετε παρακαλώ. Madame Guillaume. Κύριε Guillaume. Oui, j'avais prévu de parler de prisme, mais euh, j'ai parlé d'autre chose parce que je, je veux d'abord préciser d'entrée que je suis, personnellement, je suis très sensible et très. Ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρή με πρόσωπα ή ομάδε στη συμπεριφορά του που θεωρώ παραγωγείται κατά τον όρομα είναι κάτι σαν συλλογική μνήμη που λειτουργεί κατά τον Ρώμα, τουλάχιστον στην Γαλλία. Πέρσι έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά συνέβαλε και τότε ο πρόεδρος και ο πρόεδρος Αργοζή και επίσης κάτι σαν blackout, σαν συλλογική μνήμη γιατί είπαμε ότι έχουμε εκδιώξεις από τα στρατοπεδά τους. Αυτό σχετιζόταν με την ε, εγκατάσταση ή μη ε, αποχωρητηρίων. Σας το λέω κυρία δεν το ξέρετε, έχουμε περισσότερους από 400 οι οποίοι κρατούνται σε κάποια στρατόπεδα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε αντί για αυτό να το βοηθήσουμε στην κοινωνική του ένταξη. Κύριε Επίτροπε, έχουμε κάποιες ε, εκθέσεις που αφορούν τους Ρωμά. Και αυτές οι εκθέσεις συμφωνούν ότι είναι τα κατάσταση πάρα πολύ αρνητική όσον αφορά το τα, του σχολεία είναι ε, την ένταξή τους και όλα αυτά. Πεςτε μας επομένως, μήπως είναι δυνατόν από ε, τα λόγια να περάσουμε στα έργα και τελικά οι χώρες να μπορέσουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ. Λέω κύριε Ρωμέβα. Δύο ερωτήσεις. Για ζώμα πέραν των όσων ε, ελέγχθησαν θα πρέπει να σας ε, πω το εξή. Τι λέτε κύριε Αντιπρόεδρε για την ομάδα Μπάλατο που παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής για τους ε, Ρωμα. Πώς, πώς βλέπετε το έργο αυτής της ομάδας. Κάτι άλλο το οποίο έχει χρονίσει ως υπόθεση που εκκρεμεί. Είχα λάβει και εγώ μια έκθεση κατά των ε, δυσμένων διακρίσεων επί τη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Ε, υπήρχε υπάρξει μια εμπλοκή στο Συμβούλιο λόγω της στάσης της Γερμανίας και εμείς έχουμε απευθυνθεί στο Συμβουλίο για να ξεμπλοκάρει την κατάσταση τουλάχιστον 11 φορές. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να απεμπλακεί η υπόθεση. Πάντως σήμερα έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος της θητείας σας. Είχατε δεσμευθεί να κάνετε κάτι σε σχέση με αυτό. Πέστε μας. Μπορείτε κάτι να κάνετε παραπάνω, θέλετε κάτι εμείς να κάνουμε. Κάπως τι να γίνει, να αποσπάσουμε μια υπόσχεση από το Συμβούλιο κάτι θα γίνει. Για κολλήνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, έχω τρεις πάρα πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα. Πάρα πολύ καλά μας είπε σήμερα η κύριε Επίτροπος ε, το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων Επίσης έχουμε το θέμα των ε, φυλακών. Είναι θέμα βέβαια εθνικό, αλλά έχουμε το πρόγραμμα Στοκχόλμης, το οποίο ορίζει το ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης όταν έχουμε ε, κάποιους οι οποίοι θυγόνται προέρχονται από τρίτα, ε, τρίτες χώρες ή από άλλη χώρα. Και είπαμε ότι ένα σχετικό πρόγραμμα 2014-2020 και όσον το πρίσμα. Ακούσατε τι είπαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί ξεπέρασαν κάποια λογικά όρια αυτή τη φορά και θα πρέπει ε, να, τελικά να μπορέσει να απαντήσει ο Αμερικανός υπουργό στην Επίτροπο. Και επί τη βάση αυτών που θα πει θα πρέπει να προβληματιστούμε. Τελευταίο που θα σα αφαιρεί κύριε Πρόεδρε αφορά τον ε, Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Εγώ έχω αναλάβει μια έκθεση όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με την ε, ειδική μας ε, επιτροπή, σε σχέση με τα όσα επίσης ανέφερε και η κυρία Ρέντινγκ για τον ε, εισαγγελέα, θα πρέπει οπότε να έχουμε ένα ευέλικτο σχήμα, θα πρέπει επίσης να έχει αρμοδιότητες ξεκάθαρες η θέση αυτή, ο εισαγγελέας αυτός. Να προσέξουμε τι γίνεται με το ξέπημα του χρήματος, με τη φοροδιαφυγή, ε, μήπως και αυτά είναι αρμοδιότητες. Και έτσι επομένω να υπάρχει και έτσι μια ανάσχεση του, του οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό πρόκειται ουσιαστικά να βοηθήσει στη συνεργασία των αστυνομιών των κρατών μελών. Κάτι που είπαμε ότι θα πρέπει να, να, να, να, να, να, να Και εδώ βάζω τη γιατί σας βλέπω κάπως κουρασμένοι. Πρόεδρε. Όχι, όχι, καθόλου δεν είμαι ούτε κουρασμένος, λέει ο πρόεδρο. Απλώς ε, πιέζει ο χρόνο και θέλουν να λάβουν το λόγο και άλλοι ε, συνάδελφοι. There you go. Ε, ε, Τα πιο πολλά ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί. Δύο επιπλέον ερωτήσει, επιτρέψτε μου, σε ό,τι αφορά τι στρατηγικέ για την ένταξη των Ρωμά. Θα το συζητήσουμε σύντομα, το ξέρω, αλλά ξέρετε ότι η έκθεση προετοιμάστηκε και με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Είναι χρήσιμο να ξέρουμε πιο πολλά για τον πραγματικό αντίκτυπο και για την έλλειψη πολιτικής προθυμίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την έλλειψη του κατάλληλου περιβάλλοντος για μια σωστή εποπτεία. Συχνά αναφέρθηκε αυτό σε θέματα ενσωμάτωσης των Ρωμά. Πείτε μας, προγραμματίζετε να υποστηρίξετε τέτοιου τύπου εκθέσεις για το μέλλον. Αυτό έγινε χωρίς την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από όσο γνωρίζω. Υποβάλαμε όμως ένα πλαιτικό σχέδιο για να υποστηριχθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τέτοιου είδους ε, εποπτεία τα επόμενα χρόνια. Ένα άλλο ερώτημα για την έκθεση Ταβάρες. Το αναφέρετε κι εσείς παρά το γεγονός ότι θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια την έκθεση, υπάρχουν δύο συστάσεις, δύο προτάσεις στην έκθεση αυτή. Η πρώτη αφορά την δημιουργία ενός διαθεσμικού τριμερούς διαλόγου στο μέλλον για το τι συμβαίνει, για παρακολούθηση της κατάστασης και άλλη μια πρόταση για την δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου της Κοπενχάγης και να δοθεί και σχετική εντολή στην ΒΡΑ. Ε, πείτε μου τη γνώμη σας για τις προτάσεις αυτές. Η κυρία Φλότο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέντινγκ, θέλω να συζητήσουμε τη συνέχεια που προτίθεστε να δώσετε σε αυτά τα ζητήματα γιατί έχουμε το θέμα της ε, αξιολόγησης, γίνεται της έκθεσης του Σεπτεμβρίου όσον αφορά αυτό το παράνομο πρόγραμμα της ε, CIA που έλαβε χώρα στην Ευρώπη με συνενοχή 15 τουλάχιστον χωρών. Έχουμε περάσει από τότε ε, ένα χρόνο. Επίσης η Λιθουανία πρόκειται να λάβει την Προεδρία της Ένωσης υπ' αυτούς τους όρους. Αυτή η χώρα που κατηγορείται στα πάρα πολύ σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκθεση γιατί έχουμε αυτές τις πτήσεις και τις ε, σχετικές επιβαρυντικές αναφορές της, ε, του, του Eurocontrol. Και επίσης έχουμε την έκθεση του Μαΐου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Επίσης, τα θύματα θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή ε, και το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων απευθεία. Ούτω ώστε να έχουν ε, ελπίδε ε, ελπίδες αποζημίωσης και αποκατάσταση Έχουμε ας πούμε τις κατηγορίες κατά Πολωνία, Ρουμανία, Λιθουανία. Κύριε Αρέντι, τι πρωτοβουλίε έχετε πάρει ή θα πάρετε. Πώς επιτέλους θα σταματήσει αυτή η κάκιστη πρακτική που δηλαδή αφήνεται ξέφραγο αμπέλη την Ευρώπη να κάνουν ό,τι θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Και τώρα είδαμε τι έκανε η Εθνική Υπηρεσία ε, Ασφαλείας στην Αμερική. Τι είδους εταίρος ε, είναι αυτός. Κύριε Μομπρέ, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, πίτροπε κυρία Μορβάη. Για ε, το yes we can, για να yes we can, το σύνθημα εκείνο άλλαξε ο του κύριου Ομπάμα και τώρα τσεκάρουν τις ιδιωτικές συνομιλίες και επικοινωνίες όλων. Ακόμα και στο G8 έγινε το ίδιο. Τι θα γίνουν τα τρομερά δικαιώματα, γιατί είναι πάρα πολύ περίοδο όταν μιλούμε για προστασία ιδιωτικών δεδομένων, προσωπικών δεδομένων, Σα προβληματίζει και κολλάτε στην Ουγγαρία, στο αν έχει, αν έχει διαμεσολαβητή ή άλλου είδους ε, νομικό πρόσωπο για τα, για τα ιδιωτικά δεδομένα η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, μα μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσετε αυτού του είδους τον πόλεμο που έχετε εξαπολύσει που αντί να είναι υπερδιατλαντικό είναι ε, αντιουγγρικό αγώνα. Και έχουμε όλους τους, αυτούς τους επιφανείς, ε, εσάς δηλαδή, τον κύριο Ταβάρες, από τους οποίους μαθαίνουμε το πόσο χρειάζεται να υπάρχει διάκριση εξουσιών και δικλείδες ασφαλείας στην Ουγγαρία. Μια που είστε επομένως τόσο σημαντική κυρία, ε, πέστε μας, τι είδους συναντήσεις αυτές που είχατε, τι ελέγχθες αυτές τις συναντήσεις. Από πού προκύπτει ότι αυτέ οι μυθιαστές συναντήσει ήταν σύνομες, ήταν τέλο πάντων συνάδουν με την ελευθερία του τύπου. Τι γίνεται με, με, με, το, με το κλαμπ τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ που πάτε και τα λέτε εκεί πέρα μυστικά και δεν λέτε τίποτα. Είπατε τίποτα για την Ουγγαρία, είπατε τίποτα για τι ε, εκλογέ. Αυτό που είπε ο κ. Σόγκορ. Γιατί τα μη στην Ουγγαρία οργιάζουν με τέτοιες φήμες και δημοσιεύματα. Για, πάρτε, για, για σοβαρευτείτε. Πάρτε τα σοβαρά την υπόθεση της ε, Ουγγαρίας. Σοβαρευτείτε και απαντήστε στο σοβαρά γιατί εδώ πέρα είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σάλα Φράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αποφασιστικότητά και σα συγχαίρω. Επίση, σα συγχαίρω για την αποφασιστικότητα τη, το, το, την κατηγορηματικότητα με την οποία ε, αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όλες αυτές τις, τις, ε, τις φήμες ε, από Ουάσιγκτον και από τα Αμερικανικά ΜΜΕ και μπράβο για τον τρόπο που έχετε αντιδράσει. Επίσης, στις 14 Ιουνίου ε, προέβηται εις, ε, ε, κάποιες δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης και νομίζω ότι αφού άκουσα κάποιες αγορεύσεις Τη συζήτησή μας ότι δεν έχουν όλοι υπόψη τους το τι έγινε εκεί. Και το κύριο Ρομέρο, ε, η κυρία Ρομέρο ανέφερε κάποιον ε, ε, κάποιον χιουμορίστα, κάποιον τέλος πάντων διασκεδαστή, Ισπανό. Όμως θα πρέπει κανείς για να σατηρήσει να έχει ξαναξύρει το background. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτά τα που γίνονται στην Αμερική δεν αφορούν μόνο τους Ευρωπαίους αφορά και άλλους οι οποίοι κατηγορούνται για τρομοκρατία ή για κυβερνοκλήματα. Και η κυρία Ρέντινγκ τότε είχε πει ότι είναι αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, στον ιδιωτικό βίο είναι κυρίαρχο. Τα είπατε όλα αυτά και μπράβο. Τώρα για πέστε μας. Τι εκρεμεί και πρέπει να ξεκαθαριστεί κατά τις συναντήσεις της διατλαντικής ομάδας. Και για το TTIP πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κ. Βάνιχολτσε, να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Γιατί μιλήσαμε πολύ σε ό,τι αφορά θέματα εμπιστοσύνης μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεωρώ ότι τίθεται και θέμα ειλικρίνειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας θυμίσω μία έρευνα την οποία ανέθεσε η δική μας Επιτροπή και παρουσιάστηκε στις 20 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, για το έγκλημα Και διαπιστώθηκε λοιπόν στην έρευνα αυτή, σε ό,τι αφορά τα clouds, το υπολογιστικό νέφος ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το θέμα και θα πρέπει να κοιτάξουμε ιδιαίτερα τις ε, αμερικανικές νομοθεσίες. Αλλά δεν ε, εξαγάγαμε συμπεράσματα από όλα αυτά. Είναι νομίζω σημαντικό να προσθέσουμε εκ νέου το άρθρο 42, να το επαναφέρουμε. Συζητάμε, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, ε, μια συμφωνία εμπορική με τις ΗΠΑ. Αλλά αυτή δεν λειτουργεί. Πώς μπορούμε να συζητάμε τέτοιες συμφωνίες όσο υπάρχουν μεγάλα κομμάτια τα οποία δεν λειτουργούν. Τι συμπεράσματα θα πρέπει να εξαγάγουμε και τι σημαίνει συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Κύριε Γιάροκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα στη συνάντηση. Ήμουνα στην Επιτροπή Γυναικών και παρουσιάστηκε το έγγραφο για την αξιολόγηση ε, της στρατηγικής ε, για τους Ρωμά. Περιμένουμε την ανακοίνωσή σας και τη θέση σας για αυτά που κάνει η Γαλλία και άλλες χώρες για τους Ρωμά. Θα ήθελα να σας πω πριν, ότι πριν βγει το έγγραφο, ένα από τα μεγάλα ε, εμπόδια που θεωρούμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια είναι ότι, είναι ότι δεν υπάρχουν δείκτες, ε, βασικές γραμμές και ποσοτικοί στόχοι που θα μας επιτρέψουν να μετρήσουμε την πρόοδο. Χρειαζόμαστε τέτοιες ε, εκθέσεις από τους ίδιους τους Ρωμά που θα μας λένε πώς ε, λειτουργούν αυτά τα προγράμματα. Αλλά δεν υπάρχουν όμως ούτε κυρώσεις ούτε κίνητρα. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα, δεν θα μεταφράσουν σε καλά αποτελέσματα οι προσπάθειες. Γίνεται μαζί με σας τα εθνικά σημεία επαφής να βάλουν αυτή την ιδέα με κάποιο τρόπο στο πίνακα αποτελεσμάτων, στο scoreboard, του, ώστε να έχουμε κοινού δείχτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Είσαστε έτοιμοι να ζητήσετε ποσοτικά στοιχεία από τα, κράτα, από τα κράτη-μέλη στις εθνικές τους στρατηγικές. Προς το παρόν, μέχρι στιγμής μόνο η Ουγγαρία έχει τέτοιους στόχους γραμμένους σε χάρτου η κυρία Παπαδοπούλου, αλλά προσπαθήστε να είστε σύντομοι γιατί έχουμε ξεφύγει. Κυρία Ρέτινγκ, ε, διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και ξέρω πόσο αποφασιστικά προωθείτε την ιδέα για συμμετοχική δημοκρατία και συμμετοχή των ενεργών πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Όμως γύρω μας βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλά σοκς. Υπήρχε πρόσφατα κούραμα καταθέσεως στην Κύπρο, haircut, ουσιαστικά το δικαίωμα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την περιουσία τους και τις καταθέσεις τους έχει εκτοπιστεί, έχει παραβιαστεί. Στην Ελλάδα γίνεται παραβίαση του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Κλείνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η συμμετοχική δημοκρατία χωλαίνει. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών με όσα συμβαίνουν και ιδίως με το τελευταίο σκάνδαλο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όλα αυτά είναι σοκς. Πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Να πούμε ότι η συζήτηση αυτή απαιτεί πιο πολύ χρόνο από όλους τους συναδέλφους. Δύο μέλη από τη ΕΔΑ, η κυρία Ματιέ και η κυρία Σίπελ, ζήτησαν να ξαναμιλήσουν αν ε, δεσμευτείτε ότι θα μιλήσετε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ταβαρές, αν δεν σας είδα κύριε Ταβαρές. Λυπάμαι. Έχετε το λόγο και μετά 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, ναι, πολύ ωραία. Δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Κύριε Ταβάρες, τελευταίο παίρνετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Ταβάρες. Κύριε Αντιπρόεδρε. να επικεντρωθώ στο άρθρο 42. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στην έκθεση σήμερα. Ασφαλώς θα περιμένω να ψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Το μόνο που θα πρέπει να διευκρινίσω για την Ουγγαρία είναι για το νέο νόμο για την δημόσια ασφάλεια. Δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση και ζήτησα επίσημη μετάφραση από τις Ουγγρικές Αρχές, οι οποίες όμως δεν μου την έχουν διαβιβάσει ακόμα την επίσημη μετάφραση αυτή περιλαμβάνει πολύ ανησυχητικά στοιχεία γιατί επιτρέπει υποκλοπές επικοινωνιών και μάλιστα σε τακτική βάση για υψηλούς αξιωματόχους, δημοσίους υπαλλήλου του Ιγκρικού κράτους, μεταξύ άλλων και εισαγγελέων και δικαστών. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρό είναι για θέματα διάκρισης των εξουσιών και σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό απόρριτο, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο γενικό θέμα του άρθρου 2 του άρθρου 2, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα, μια ομάδα αξιών που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν απαραίτητα. Θα χρειαστεί πολιτική απόφαση και έλεγχος προκειμένου σωστά να εφαρμοστούν. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να δημιουργηθεί η ομάδα υψηλού επίπεδου της Κοπεχάγης όπως διευκρινίστηκε. Θεωρώ ότι η ατζέντα αυτή θα συνάδει σε όλα όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω για τις δικές σας απόψεις επ' αυτού και σε ό,τι αφορά και την ομάδα υψηλού επιχειπέδου της Κοπενχάγης. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σας παρακαλώ, συνάδελφοι, παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία γιατί θα μιλήσει η Επίτροπος. Θα μιλήσει η Επίτροπος για να απαντήσει στα ερωτήματα που της ετέθησαν. Θα, θα χρειαστεί κάποια λεφτά, αλλά σας παρακαλώ πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και αυτό καταδεικνύεται από τον υψηλό αριθμό συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Έχετε το λόγο, Επιτροπέ. Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθούν όλα αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα, τα οποία πραγματικά χρειάζονται πιο πολύ χρόνο και πιο ενδελεχείς απαντήσεις. Αλλά ξέρω ότι σε κάποια από τα θέματα αυτά θα επανέλθουμε όταν το Κοινοβούλιο θα υποβάλει τις προτάσεις του. Τώρα, για να απαντήσω εν συντομία σε ένα από τα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ε, σύνοδο αυτή. Bildenberg. Να σας απαντήσω εντάχει. Όλα αυτά δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με την πραγματικότητα σε καμία έκφανσή της. Τώρα, να περάσουμε στα πιο σοβαρά πράγματα. Το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Συμφωνώ με όλους τους βουλευτές που ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει ο κανονισμός και η οδηγία να παραμείνουν μαζί, ενωμένα. Συμφωνώ και με όσους είπαν ότι υπάρχει μια, ένα απαράβατο όριο, ένα συνεκβανόν. Τα δικαιώματα της οδηγίας του 95. Δεν θα συνενέσω σε καμία περίπτωση να μην τηρηθούν αυτά τα δικαιώματα και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα του οίκου μας σε πρώτη φάση, σε τάξη. Σίγουρα αυτό είναι ένα μέρος της απάντησης που μπορούμε να δώσουμε προς τους Αμερικανούς εταίρους μας. Για μας είναι κατεπήγον το θέμα αυτό θα πρέπει οι δικοί μας οι κανόνες να είναι ξεκάθαροι. Γιατί αυτό θα συνεπαγόταν επίσης ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εθνικότητος, ανεξαρτήτως τοποθεσίας της μητρικής εταιρείας ανεξαρτήτως ε, της έδρας, της τεχνολογικής έδρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά ύψιστη σημασία. Πού βρισκόμαστε τώρα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και τη σχετική μεταρρύθμιση. Δεν ε, θα συζητήσω το ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αυτό το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από όλους. Με ρωτήσατε όμως τι γίνεται στο Συμβούλιο. Είναι πολύ αντικρουόμενα, αν θέλετε, και περίεργα τα μηνύματα τα οποία δίδονται για το τι έχει συμβεί de facto στο Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία, η οποία και έκανε εκπληκτική δουλειά. Κατάφερε να επικεντρωθεί στο κεφάλαιο 1-4 του κανονισμού και έχει θέσει επιτάπητος αναθεωρημένο σχέδιο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο τα έχει επικροτήσει αυτά. Παρά το γεγονό ότι, ήταν μικρή η μειονότητα ότι υπήρχε μια μικρή μειονότητα κρατών που προσπάθησε να μπλοκάρει τα πράγματα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία τα ενέκρινε. Για την οδηγία, η πρώτη ανάγνωση έχει ολοκληρωθεί στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο λοιπόν προχωρά. Καλά μάλιστα και είμαι αισιόδοξη θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μετά ιδιαίτερα από την υπόθεση Prism, θα συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε προτού ε, πριν τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου θα ληφθούν οι αποφάσεις. Τώρα, για την υπόθεση Prism. Αληθεύει, στέκει ότι απέστειλα επιστολή στις 10 Ιουνίου στον Eric Holder για να ζητήσω να απαντηθούν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όντως, κάποιες από τις ερωτήσεις απαντήθηκαν στην συνάντησή μας στην Ιρλανδία. Επίσης, αληθεύει ότι δεν απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα. Και γι' αυτό ο συνάδελφος, η συνάδελφος Μάλμστρομ και εγώ αποστήλαμε μια επιστολή εκ νέου προς τον Γενικό Εισαγγελέα αναφέροντα τα εξή. Στη συνάντησή μα δεν ήμασταν ακόμα σε θέση να απαντήσουμε όλε τι ερωτήσει που ετέθησαν στην επιστολή τη 10η Ιουνίου και δεδομένη τη κοινή γνώμη και τη ε, περίεργη στάση που τη περίεργη διάθεση που επικρατεί από την πλευρά μα του Ατλαντικού, θα θέλαμε να απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν τα ερωτήματα αυτά και μα ανησυχούν ιδιαίτερα ο όγκο των ε, δεδομένων που συλλέχθησαν και η ο σκοπός του πεδίου εφαρμογή του προγράμματος και οι δικαστικές οδοί και οι συλλογικές δικαστικές οδοί που διατίθενται, έχουν δυνατότητα να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή λοιπόν είναι Αυτέ είναι οι ερωτήσει και εγώ και η Σεσίλια ζητήσαμε να ξεκινήσουν οι συναντήσει αυτέ τον Ιούλιο. Να μην αναπευθούν στι ελληνικές καλένδε λοιπόν αυτά, αλλά να είναι άμεση η αντιμετώπιση τους και να υπάρξει απάντηση στην επιστολή μας πριν ξεκινήσουν οι συναντήσεις της ομάδας. Αυτά λοιπόν ως εδώ. Και ναι, η δήλωση που έκανα μετά την συνάντηση με τον Eric Holder αποτελεί την επίσημη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Ελπίζω, Πρόεδρος, ελπίζω, Πρόεδρε, όλα τα μέλη της Επιτροπής να λάβουν την επίσημη δήλωση. Τώρα για τα διάφορα τέτοια ζητήματα που Ακούσαμε τις διάφορες ερωτήσεις για, την... για τους κανόνες των προσωπικών δεδομένων και προστασία των προσωπικών δεδομένων και πώς αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι πριν από 18 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε μία, έκανε μία πρόταση και η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάλλον αυτή ήταν η επίσημη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ήταν οι προηγούμενες ε, προτάσεις που είχαν μορφή σχεδίου. Τώρα, ετέθησε μια συγκεκριμένη ερώτηση για ένα άρθρο, το άρθρο 42, όπως το αποκαλείται. Αν διαβάσετε την ιδεολογική σκέψη 90, θα δείτε ότι περιλαμβάνεται στο σχέδιο κανονισμού. Με μεγάλη σαφήνεια. Οι αρχές επιβολής του δικαίου σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ζητήσουν πληροφορίες μέσω νόμιμων διόδων. Νόμιμες δίωδοι ποιες είναι. Ξέρω ότι στο κοινοβούλιο αυτό έχουν κρατηθεί σχετικές τροπολογίες προκειμένου να γίνει η τελογική σκέψη αυτή ένα άρθρο του διστακτικού. Θα ζητήσω από το Κοινοβούλιο να λάβει τι ευθύνε του. Αν θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει η τελογική σκέψη να μπει στο διδακτικό, εντάξει, εγώ δεν έχω οποιαδήποτε αντίρρηση. Θα ήθελα να πω ότι το Patriot Act από το 2011 σε όλες τις συναντήσεις με τους Αμερικανούς έχει τεθεί επιτάπητος. Γιατί, επειδή αν πάει κανείς κατευθείαν στις ε, επιχειρήσεις και ζητά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, αυτό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό διαρκώς επαναλαμβάνεται και αυτό αποτυπώνεται στο, στην ιδεολογική σκέψη 90. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για θέματα μυστικών υπηρεσιών, πληροφοριών. Φυσικά, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι εντός της δικαιοδοσίας μας. Ε, κοιτώντας όμως ε, τις δηλώσεις που έγιναν, αναφέρεται ότι ακόμα και σε θέματα τέτοιων πληροφοριών, τέτοιων μυστικών υπηρεσιών, οι βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο κείμενό μας δεν παραγνωρίζονται. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άρα η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται χωρίς οποιαδήποτε σκιά και χωρίς οποιαδήποτε υποψία αμφιβολίας. Κάτι άλλο τώρα. Το πακέτο για τα διαδικαστικά. τα δικονομικά δικαιώματα. Όπως είπα, ε, στην εισαγωγική μου παρουσίαση έχει δρομολογηθεί και εμπεριέχεται και η νομική βοήθεια στο εσωτερικό του πακέτου, όπως σας υποσχέθηκα πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξεκαθάρισε επίσης το ίδιο και στο Συμβούλιο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πρόσβαση σε δικηγόρο. Κάτι που συμφωνήθηκε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτή την πρόσβαση σε δικηγόρο. Τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη νομική βοήθεια. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους ευπαθείς ε, υπόπτους και για το τεκμήριο της αθότητας. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν το φθινόπωρο, θα έχετε όλα αυτά τα θέματα επιτάπητος. Πρόεδρε, ούτως ώστε να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε όταν επιστρέψετε τις διακοπές. Το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων που πετούνται ασύλου είναι ένα θέμα της Σεσίλια. Προσπαθώ να είμαι να τον πιο λακωνική. Αν δεν απαντήσω όμως με κατηγορούν τα μέλη της Επιτροπής σας ότι δεν απαντάω. Με την ησυχία σας λέει ο Πρόεδρος. Άρθρο 19. Το 19, η οδηγία στο άρθρο 19, μιλάμε για την οδηγία του 2008, το άρθρο αυτό είναι μπλοκαρισμένο. Κάθε Προεδρία προσπαθεί να το απεμπλέξει, αλλά κάθε φορά έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Όταν ταξιδεύει κανείς στα κράτη-μέλη, ξέρετε πολύ καλά ότι τότε φαίνεται πως δεν είναι ένα κρατός μέλος που μπλοκάρει το θέμα, αλλά μια ομάδα κρατών μελών. Επιπλέον η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία και επομένως έχουμε αυτή τη θέση στο Συμβούλιο. Το μπλοκάρισμα αυτό στο Συμβούλιο. Εμείς δεν αποσύρουμε αυτή την πρόταση. Είναι θέμα αρχής. Είναι καλή η πρόταση. Και η πλειοψηφία, η ευρεία πλειοψηφία των κρατών μελών την υποστηρίζει την οδηγία αυτή. Γιατί να την καταστρέψω λοιπόν. Όχι, θα, θα παραμείνει. Η Κομισιόν δεν χρειάζεται να επαναχωρήσει από μια θέση που βρίσκεται σύμφωνο το Κοινοβούλιο και την πλειοψηφία των κρατών μελών, μόνο και μόνο γιατί μια μειοψηφία κρατών μελών μπλοκάρει αυτή την πρόταση. Εγώ κάθε Προεδρία την ενθαρρύνω να συνεχίσει τι συζητήσει και να επιδιώξει το συμβασμό για τους Ρωμά. Έχουμε ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011, ε, επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι μόνο από το Συμβούλιο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και τα κράτη-μέλη παρουσίασαν τις εθνικές στρατηγικές τους για την ένταξη των Ρώμα. Πρέπει αυτή την ορμή που έχει δημιουργηθεί να την κρατήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε και πιο μπροστά. Θα το κάνουμε αυτό πώς, την επόμενη εβδομάδα, με μια πρόταση για μια σύσταση του Συμβουλίου που να βασίζεται σε μέτρα κατά των διακρίσεων. Ε, είναι νομική βάση αυτή για αυτή τη εξέταση του Συμβουλίου για έλλειψη διακρίσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση και τη σύσταση του Συμβουλίου, δύο κείμενα δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο αποτιμούμε την κατάσταση και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν φυσικά περισσότερα πράγματα και όλοι συνιστούμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν χρηματοδότης που δεν χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιήσουν πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως η εμπλοκή των τοπικών αρχών, της τοπικής διοίκησης και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, κάνουν μηχανισμούς, να έχουν μηχανισμούς παρακολούθησης και να μετρούν με αυτό τρόπο την πρόοδο αν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Στρατηγική για τους ομοφιλόφιλους, άντρες και γυναίκες, έχουμε έναν οδικό χάρτη στην Κομισιόν. Ε, οργανώνεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, νομοθετική πρόταση και πρωτοβουλίες για την ίση μεταχείριση, την έλλειψη διακρίσεων που ε, ελέγχεται με βάση το χάρτη πριν υιοθετηθεί από την Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη η οδηγία των προποθέσεων. Ε, υπήρξε ανάσχεση εδώ στον τομέα του ασύλου, πολύ συγκεκριμένα γιατί γιατί θα δημιουργούσε ε, διακρίσεις ε, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα βάλουμε το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και μόνο τότε η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, ελέγχουμε κάθε στοιχείο της νομοθεσίας που προτείνει η Κομισιόν. Δεύτερον, η Κομισιόν προτείνει και μάχεται για την νομοθεσία, να την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Η πρόταση της Κομισιόν του 2008 μας βοήθησε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ασχολείται με τις ομοφοβικές τάσεις στο ποδόσφαιρο και δήλωσε ότι αυτές οι δηλώσεις, οι ομοφοβικές, είναι διακρίσεις. Για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου έχουμε παραπέμψει κράτη-μέλη στο δικαστήριο, τη Μάλτα, Φερρυπίν, εκεί παρενέβημαν και η Μάλτα άλλαξε την εθνική της νομοθεσία, ούτως ώστε να γίνει συμβατεί με την ελεύθερη κυκλοφορία και με την έλλειψη διακρίσεων. Στον τομέα της πολιτικής, ξέρετε πολύ καλά ότι παρεμβαίνω κάθε φορά που κάτι πάει στραβά και ξέρετε ότι βοηθάμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους, να προωθήσουν ίδια δικαιώματα για τους ομοφιλόφιλους και τους φιλομεταβατικούς στην Ευρώπη. Ε, πίνακας επιδόσεων για τη δικαιοσύνη. Ο πίνακας αυτός αποτελεσμάτων ή επιδόσεων έχει μπει στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εγώ δεν περίμενα θα τα καταφέρουμε. Αλλά πέρασε. Και τώρα. Με βάση αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων, 10 χώρες έφτιαξαν τις συστάσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τις δεχτεί για να δούμε αν θα το κάνει να θα τις δεχτεί αυτές τις συστάσεις. Γιατί αν το κάνει, αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Συμφωνώ όμως με αυτούς που λένε ότι αυτό δεν λύνει το βασικό θέμα του κράτους δικαίου. Το άρθρο 7, ατομικά όπλα και το δίλημα της Κοπενχάγης. Το δίλημα της Κοπενχάγης. Τι θα κάνουμε, γιατί μάλλον δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 7. Το συζήτησε το Συμβούλιο. Το Τζάι τον Ιούνιο, το ΓΚΑΤ τον Απρίλιο. Θα γίνει και άλλη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και θα γίνει και άλλη μια συνεδρίαση τον Αύγουστο του Συμβουλίου αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Θέλουμε να, το, να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για την άποψη της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει στην Ολομέλεια το θέμα αυτό και τον Νοέμβριο θα γίνει το Assis de la Justice. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία δεν έχει να κάνει με τα επιμέρους προβλήματα που θέλουμε να επιλύσουμε. Μιλάμε για την οριζόντια λύση που πρέπει να εφαρμόσουμε κάθε φορά που θέλουμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο. Ξεκαθάρισα ήδη στο Συμβούλιο και θα το ξεκαθαρίσω και σε εσά ότι πιστεύω πως η καλύτερη λύση είναι κάτι που να μοιάζει με το άρθρο 121 που προβλέπει τα κάποια οικονομικά και ρυθμίζει οικονομικά ζητήματα. Αλλά αυτό θα απαιτήσει αλλαγή τη συμφωνία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναλύσουμε και εμεί και όλα τα θεσμικά όργανα για να δούμε με βάση τι σημερινέ συνθήκε τι, έχ, λύσεις έχουμε και ποιες ε, είναι οι βέλτιστες λύσει για πιθανή αλλαγή τη συνθήκε. Άκουσα και είδα τι έγραψε ο κ. Σταβάρη στην έκθεσή του και αν συμφωνήσει με την έκθεσή του η Ολομέλεια θα διοργανωθεί μια ομάδα υψηλού επίπεδου Κοπενχά... ομάδα Κοπενχάγης και θα είναι αυτή μία από τις δράσεις που θα προωθήσουμε. Θα περιμένουμε όμως και την απόφαση ε, της Ολομέλειας. Το θέμα του κ. Ταμβάρης για τον Ουγγρικό νόμο για την επιτήρηση. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο ανησυχεί για αυτή την νομοθεσία, αλλά πριν κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να αναλύσουμε την νομοθεσία. Όταν η Κομισιόν κάνει μια ανάλυση και προβαίνει σε πρόταση, ε, λειτουργεί σαν δικαστικό σώμα. Επομένως, θα πρέπει η ανάλυση μας αυτή να είναι πολύ ενδελεχής. Για το θέμα της Βουλγαρίας, ελπίζω πρώτον η Βουλγαρία να τα καταφέρει να περάσει σε διαρκείς μεταρρυθμίσεις και δεύτερον, σημείωσα ποιο είναι ο υποψήφιο που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, ο οποίο αποσύρθηκε και ελπίζω τελικά ο πρόεδρο ε, όταν διορίσει τον επόμενο να υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία. Κυρία Φλότρον, για τις μυστικές κρατήσεις και απαγωγές της CIA με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου εγώ και η κυρία Μάτσομ στις αρχές του 2013 στείλαμε μια επιστολή σε όλα τα κράτη-μέλη όπου θέτουμε δύο βασικά ερωτήματα. Τι μπορεί να γίνει για να ανακαλύψουμε την αλήθεια και τι μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη. Έλαβα όμως λίγες απαντήσεις. Πολύ μακροσκελή ήταν η απάντηση, δεν είναι συνηθισμένο αυτό, αλλά καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητερα είναι τα θέματα που, στα οποία απάντησε η Επίτροπος. Σας ευχαριστώ για την ε, υπομονή σας. Έχουμε καθυστερήσει για τις ψηφοφορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο που κατάφερε να απαντήσει και στα 30 μέλη της Επιτροπής μας που ζήτησαν το λόγο και έκαναν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Τα κατάφερε να τους απαντήσει. Okay, now... Πρόεδρος. Λοιπόν, έχετε τις κάρτες για την ψηφοφορία, τις ηλεκτρονικές κάρτες. Πηγαίνετε να τις πάρετε ή στείλετε κάποιον στις φέρει, εντάξει, για να ψηφίσουμε. Okay, let's catch up. Proceeding to the vote. Every member. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Shall we still take a minute, minute of recess? Do you... Θέλετε δύο λεφτάκια διάλειμμα, κυρία Ματιέ.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 Shall we go? Να ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Το έλκα, έτοιμο. Θέλετε άλλα δύο λεπτά. di tempo. Shall we go? Shall we go? Να αρχίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. We're voting on the right of access to a law. Θα πρέπει να ψήσουμε τώρα το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Δεύτερη ψηφοφορία για σήμερα και αρχίζουμε με όλο μαζί το κείμενο που απαιτέλεσε αντικείμενο συμβασμού. Έτσι δεν είναι, να κατάλαβα καλά. Εάν τηρήσουμε το συμβαστικό κείμενο, αυτό που συμφωνήθηκε κατά μόνο μια ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές. Ωραία, επομένω εγκρίνεται, εντάξει. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. What do we see? 49 plus. 49 υπέρ. 2 κατά. Καμία αποχή. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια κυρία Αντωνέσκου. Προχωρούμε τώρα. Ποιο ηγητή το λόγο. Α, η κυρία Αντωνέσκου. Έχετε το λόγο. Știu că foarte prost cu uh, timpul, de aceea o să uh, fiu foarte scurtă, dar nu... Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο. Πρέπει να ευχαριστήσω του συναδέλφου. Ήταν ομαδική, συλλογική η προσπάθειά μα, Βοήθησαν και σκιώδες ηγητέ. Δεν θέλω κανένα, από κανένα θέλει να αστερίσω τη, τη, για την επιτυχία, αλλά ευχαριστώ και την ε, ε, κυρία Ρέντινγκ, επίσης τους συνεργάτες των πολιτικών ομάδων, ε, οι συνεργάτες μας και φυσικά κυρίως οι γραμματεία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ όλους. Και, Ρομέρο. Τι συμβαίνει κύριε Ρομέρο. Κυρία Ρομέρο. δήλωση σε σχέση με την ε, ψηφοφορία. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ψηφίσαμε υπέρ. Γιατί βελτιώθηκε η κατάσταση, βελτιώθηκε το κείμενο. Πάντω, ω πολιτική ομάδα δεν συμφωνούμε με κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτό δηλαδή που αφορά του λόγου για τη σχετική εξαίρεση όσον αφορά λοιπόν την αποστέρηση κάποιου του δικαιώματος πρόσβαση σε δικηγόρο επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε για το θέμα αυτό ή στο μέλλον. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ε, θα ελήφθη υπόψη η δήλωση η επεξήγηση της ψήφου τέλος πάντων και τώρα θα εληφθη υποψη η δηλωση η επεξηγηση τη ψηφου τελο παντων και τωρα θα προχωρησουμε η στην επόμενη ψηφοφορία είναι το κείμενο του κυρίου Μίλντερ. Πρόκειται για την έκθεσή του που αφορά την θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος επιτήρηση των Συνόρων. Αυτό δεν είναι. Και θα κάνουμε το ίδιο όπω και πριν. Έχουμε ένα συμβαστικό κείμενο ε, θα ψηφίσουν όλα μαζί επομένως και εδώ με ηλεκτρονικός έλεγχος ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά άποχες εγκρίθηκε και τώρα ηλεκτρονικός έλεγχος τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρας 41 υπέρ, 8 κατά, μία εποχή. Ευχαριστούμε κύριε Μίλτερ για το ε, ενιαίο συμβαστικό κείμενο. Και τώρα προχωρούμε. Έχουμε και κάποιες άλλες ψηφορίες ε, και κάποιες ε, τροπολογίες. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματο όσον αφορά την εφαρμογή τη στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Let's start with the voting. Amendment 1. Those in favor. Πρώτη τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ε, πρέπει να γίνει έλεγχος. Let's have a check. Okay. Adopted. Thank you. Now, amendment. Εγκρίνεται τώρα η τροπολογία παραθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία παραθμών 3 υπέρ για το 3 κατά αποχές συγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται. Έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκρίνεται. Εφτά. Υπέρ. Κατά. Mm. Seven. The vote is open. Για ε, το 7 ψηφίζουμε. Α, εδώ πέρα αυτό. Υπάρχει κάποια διαχωριστική γραμμή. Μ, βλέπω, βλέπω. 31 19. κατά 19. Σαφώς είναι και τροπολογία τώρα υπερθυμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά δεν σήκωσαν αρκετοί το χέρι ιδίω ε, στη μέση της αιθούσης θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο για το 12 ψηφίζουμε πέρας 34 κατά 17. Α, είναι θέμα του πώς σήκωσαν το χέρι. Δεν είναι, δεν είναι αριθμοί, είναι τα χέρια. Now, moving on, 11. Πάμε τώρα στο 11. Υπέρ, κατά αποχές. Απο, 13, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 14, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Λειτουργικός έλεγχος για το 14. πέρας. Νομίζω ότι απολύτω πρέπει να κάνουμε καταμέτρηση. Γιατί ιδίω ε, υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικέ ομάδε που δεν έχουν σηκώσει αρκετοί από αυτέ τα χέρια. Τι θέλετε κύριε κυρία θέλετε λόγο. Ε, ε ψήφισα λάθο προηγουμένω. Λάθο λέει ο πρόεδρο. Υποθέτω ότι ηλεκτρονικά θα το διορθώσουμε. Να δοθούν οδηγίες, ώστε να γίνει ηλεκτρονική διόρθωση. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το 18 έχει αποσυρθεί. 16. Με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 22 προφορική τροπολογία, συγγνώμη, 21, 21 διορθώνει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 22 προφορική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25. 22. Θα κάνουμε για το 22 ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. 22-28. Απορρίφθηκε. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ όχι τι συμβαίνει έλεγχος για το 28 Πέρασε. Εγκρίθηκε. 30. Υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Α. Α, όχι, όχι, καταπίπτει το. 32. Όχι και το 32 καταπίπτει. Όχι. Καταπίπτει ή όχι. Το 32 δεν καταπίπτει ισχύει. Επομένω πρέπει να το ψηφίσουμε. 32 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Διεθνικός έλεγχο για το 32. Πέρας. 20 το 7-23 εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια σας. Μερικές πολιτικές ομάδες βαριούνται περισσότερο από άλλες και δεν μπορούν να καταλάβουν τι, τι, τι, πώς διαμορφώνουν την ψήφος. 32 υπέρ. 33 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά Αποχές ε, εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Νομίζω εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Συμφωνείτε. Ναι. Το 42. Εδώ θα πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Έτσι δεν είναι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές λοιπά, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 Για να κάνουμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο για το 47. 32-20. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές Απολύτω. 55 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά θα κάνουμε τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. «25 8 με 19 αποχές. Πάντως εγκρίνεται. Δεν λέω συγχαρητήρια γιατί εγώ ήμουνα ο εισηγητής. Πάμε στο επόμενο σημείο τώρα, το οποίο ήταν το σχέδιο ψηφίσματος για την διασυνολογική συνεργασία στην εφαρμογή του νόμου απόφαση πριν και το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών. Πρώτη τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Δεύτερη τροπολογία. Υπέρ, κατά. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. 50 κατά 2. Μη 0 αποχές. Και αυτή ήταν η δική μου έκθεση, οπότε πάλι τελείωσε χαρακτήρια και πάμε στο επόμενο σημείο της Ναταλή Γκρίσμπεκ. Σχέδιο εκθέσεως για τους ασυνοδεύτους ανηλίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γκρίσμπεκ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κατέθεσα μια τροπολογία. Τροπολογία προφορική για τη δική μου, την υπαριθμόν 43. Προσθέτουμε εδώ μια νέα παραγραφό για να υπάρχει περισσότερη ιστορική συνέπεια. Αντικαθιστούμε το τέλος της φράσης και λέει για να προστατεύσουμε τους ασυνόδευτους ανηλίκους και να τηρηθούν πλήρως, να γίνουν σεβαστά απολύτως τα θεμελιώδη τους δικαιώματα.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 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γυναικών ε, διάταξη υπαριθμόν 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, διάταξη 4, Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά εγκρίνεται. Γυναικών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυναικών διάταξη 6 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Και υπερθυμών 7 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές Υπέρ, υπέρ, υπέρ για το 14. Για να δούμε. Σηκώστε ευκρινώς τα χέρια σας. Βλέπω το ΕΛΚ. Ρίζει με ξεκάθαρο τρόπο. Κατά, κατά όλοι οι άλλοι. Επομένω απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εδώ είμαστε διηρημένοι. Επί του 20. Έλεγχος επί του 20. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική παρθμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στο 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί πηδήξαμε την 27. από εδώ μέσα τρυπωμένη είναι άρνατη. Ποιοι είναι υπέρ του. 27 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβαστική. Ε, ε όχι, όχι, μισό λεπτό. Βέβαια 18 τη συμβαστική πήγαμε στο 31, 36 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, γυναικών 4 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, γυναικών 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γυναικών 15 περκατά για να κάνουμε καλύτερα έλεγχο έλεγχος για την υπαρχόν 15 γυναικών πέρασε σε 23 εγκρίνεται συμβαστική παρθμόν 3 υπέρ Κατά εποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 με προφορική τροπολογία. 43 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 46. Κατά εποχές απορρίπτεται. Δεύε 2 υπέρ. 2, 3, ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Και 8. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Αποχές. 51. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Γυναικών. Λοιπόν, 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Εδώ όμως έχουμε χωριστή ψηφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τρίτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε. Ντεβε 10. Όχι. Πάμε στην τροπολογία παριθμών 60 υπέρ. Υπέρ, κατά. κατά. Αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται 68 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 66. Ψηφίζουμε. Πέρας. 36 υπέρ, 16 κατά, υιοθετείτε. 68 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε τώρα. Θέλετε να την ελέγξουμε. Την ελέγχουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. 32 υπέρ, 30... 22 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ, υιοθετείτε. DV1 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε. ΦΑΜ 24 20... υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 8 Υιοθετείτε. Ντεβε 3. Όχι, καλύπτεται από τον συμβασμό 8. Καταπέπτει το όλο πακέτο. Πάμε στην 76. Τροπολογία υπέρ, 76 ε, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 82 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 63 υπέρ. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 5, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 9, υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. Όχι, οθετείτε, συγγνώμη. Δεύτερο πρώτο τμήμα. Ελέγχουμε την συμβαστική 9, την ελέγχουμε. Ψηφίζουμε τώρα. 30 υπέρ, 22 κατά, υιοθετείται. ΔΕΒ 7, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές υιοθετείται. ΦΑΜ 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΦΑΜ 25, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90, κατά, υπέρ, κατά, 90 με 93 τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Πάμε. Στην 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε, Συμβασμός 20. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φάμε 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ ποιο είναι το πρόβλημα θέλετε χωριστή ψηφοφορία Κύριε Αλμάιερ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Προφορική τροπολογία. Ε, και έχουμε και χωριστή ψηφοφορία εξάλλου. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα του κειμένου. Όχι το δεύτερο τμήμα. Ε, λυπάται που η τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες για την ε, υποδοχή των ε, τούντων άστων δεν απαγορεύει την κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ε, ζητάμε να ψηφιστεί αυτή η φράση, παρακαλώ. Το ΕΛΚ ζητάει αυτό το πράγμα. Θέλει χωριστή ψηφοφορία. Πρέπει να ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Ράισπεκ. Τι γνώμη έχει. Πρόεδρε, είναι πολύ αργά να καταθέσετε τέτοιο αίτημα για χωριστή ψηφοφορία. Πάνω το έχετε κάνει χθε το βράδυ. Σωστά δεν τα λέω. Είναι προφορική τροπολογία, τη διαπραγματευθήκαμε τους και δεν είναι ατελή. Αν δεν απατώμε, λέει ο πρόεδρος, για να έχουμε προφορική τροπολογία εκτός προθεσμίας, όπως στην προκειμένη περίπτωση, χρειάζεται να έχουμε ομοφωνία στην Επιτροπή. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις διαδικαστικής φύσεως, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι δική μου τροπολογία αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την αντίρρησή μου στην προφορική τροπολογία. Νομίζω ότι η τροπολογία είναι συμβατή με αυτά που ψηφίσαμε μέχρι τώρα. Ζητάμε απλώς το πακέτο ασύλου, όπως ψηφίστηκε, να επιτρέπει να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για τους ανηλίκους. Και αυτό επιτυγχάνουμε εδώ. Σεβόμαστε τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ορίζονται από την οδηγία. Τίποτα παραπάνω, επομένω έχω αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ε, ζητώ συγγνώμη, κυρία Κορέτσα Μπίλτ. Συμφώνησα με την κυρία Γκρίνσπιχ, την εισηγήτρια, που είπε ότι συμφωνούσε. Και το έχω και γραπτό μα αυτό από τη γραμματεία, ότι θα μπορούσαμε να καταθέσουμε προφορική τροπολογία για αυτό το σημείο το σημείο που λέει ε, ζητάει να συμμορφωθεί χωρίς να ξεχνάει τις ε, α, θεμελιώδεις υποχρεώσεις να μην θέτει σε κράτηση τον ανήλικο. Και ζητάει να, από τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις εξαιρετικές συνθήκες. Και το άλλο κομμάτι, διπλός μέχρι το asylum seekers, είναι χωριστό τμήμα. Ε, συμφώνησε και η γραμματεία, γιατί είναι αίτημα του ΕΛΚ. Το έχουμε και γραπτό σε αυτό, το ότι συμφώνησε η γραμματεία. Εντάξει, Κυρία Μπίλτ, καταλάβαμε τι θέλετε. Αν δεν μου τα λένε λάθος, τα του καταστατικού, οι προφορικές τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν εδώ, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτή δεν είναι όμως ε, μόνο προφορική τροπολογία, είναι μαζί και χωριστή τροπολογία. Θέλετε να χωρίσουμε την ψηφοφορία διαφορών τροπολογιών. Για να το κάνετε αυτό, για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να γίνει εν ευθέτω χρόνο. Αλλιώ θα πρέπει να υπάρχει συνένεση εδώ. Ομοφωνία δηλαδή. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ομοφωνία εδώ. Υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει. Έχετε αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. υπάρχει. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Γιατί υπάρχουν αντιρρήσει. Να ψηφίσουμε την 105 αν δεν ε, έχετε αντίρρηση. Εντάξει. Υπέρ της 105. Κατά. Αποχές. Διοθετείτε. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 107 υπέρ. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Α, μπερδεύτηκα. 108. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Και τώρα ΦΑΜ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 14 όχι 13 διορθώνει ο πρόεδρο. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. ΔΕΒΕΞ υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Φαμ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φαμ 18 υπέρ. κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 21 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Πάμε στην 155. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 157 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 161 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 164 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 167 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 168 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται φαμ 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβάσμα 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται Συμβάσμα 15 υπέρ κατά αυτές υιοθετείτε. 181 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Φάμ 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. Φαμ 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά Εποχές απορρίπτεται. 187. «184». Υπάρχει ακόμα 184. 184. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Εποχές υιοθετείται. 185. Όχι, 187. Ψηφίζουμε 187. Υπέρ. Κατά. Εποχές υιοθετείται. Συμβασμός 16. Υπέρ. Κατά. Εποχές υιοθετείται. Σεβα... Συμβασμός 17. Υπάρχει ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Συμβασμός 17 καταρχήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τώρα, το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο δεν καταπίπτει. Ψηφίζουμε το δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα. 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαν 12 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. ΦΑΜ 20 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές, το ελέγχουμε. Ελέγχουμε το ΦΑΜ 20. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 κατά 29, 22 υπέρ, 29 κατά απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 καταπίπτει. «207 υπέρ, όχι δεν καταπίπτει». «Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται». «208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». 210 υπέρ κατά Πάμε στην ε, τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρα της ψηφοφορία. 48 υπέρ. 4 ψήφοι κατά. Καμία αποχή. Κύριε Γκρίνσμπερg. Συγχαρητήρια. Now,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 It's actually 15 minutes because we... 15 λεπτά, γιατί έχουμε καθυστερήσει για να ακούσουμε μία έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τρίτη εξαμενή έκθεση για το λειτουργία του χώρου Σέγγεν στην περίοδο του από 1η Νοεμβρίου 2012 έως, 12, έως 30 Απριλίου 2013. Με την πρώτη και τη δεύτερη έκθεση καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει την έκθεση στην Επιτροπή μας σε μια πολύ συνοπτική επισκόπηση και πάλι λοιπόν τώρα έχουμε μαζί μας τα κρατημέλη και ύστερα θα δώσουμε το λόγο σε κάποιους βουλευτές αν θέλουν για να, πάρουν, να κάνουν σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την τρίτη ε, έκθεση η οποία καλύπτει από 1η του 2012 μέχρι 34 του 2013. Πρόκειται για μία διετή έκθεση και είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τον χώρο Σέγγεν. Το συζητήσατε και στην Ολομέλεια το θέμα αυτό. Χαιρόμαστε που θα μπορέσουμε σύμπτωμα να εφαρμόσουμε τον καινούριο μηχανισμό. Χαιρόμαστε επίσης που διαπιστώνουμε ότι η πίεση στα εξωτερικά σύνορα έχει μειωθεί κατά την περίοδο έρευνας ε, στα σύνορα με την Ελλάδα και την Τουρκία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε σε κάποιες περιπτώσεις ε, και τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και τα χερσαία σύνορα της Βουλγαρίας. Επίσης η κατάσταση στην Συρία προκαλεί μεγάλες ανησυχίες. Προφανώς υπάρχουν ε, ε, εξελίξεις και η κρίση τα τελευταία δύο χρόνια, αν και θα πρέπει να δηλώσουμε ότι ο αριθμός σύρων που έχει εντοπιστεί στα εξωτερικά σύνορα έχει μειωθεί. Εκ παραλλήλου, Προφανώς θα πρέπει να φροντίσουμε και να κοιτάξουμε την κατάσταση στην Μεσόγειο εν γέννη. Επίσης σημειώνουμε με χαρά ότι υπερψήφισε την ανάπτυξη του Eurosur πριν από λίγα λεπτά και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοιες ε, τραγικές περιπτώσεις. Επίσης η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Παρουσίασα τους κανόνες για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Ξέραμε ότι αυτό ήταν απαραίτητο λόγω της κατάργησης της προηγούμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν σαφείς κανονισμοί για τις επιχειρήσεις Frontex και σε ό,τι αφορά τα άτομα που ζητούν Προσβλέπουμε και στις μελλοντικές συζητήσεις με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος χωρίς καθυστερήσεις. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση εντός του Σέγγεν, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις δευτερογενείς κινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τους εμπειρογνώμονες και το Frontex προετοιμάζει ένα πλειοτικό σχέδιο για να συλλέξει τέτοιες πληροφορίες για τις δευτερογενείς μετακινήσεις και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα στις αρχές του 2014. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μοντικών πολιτικών σε σχέση με τη μετανάστευση. Επίσης, ε, πολύ σημαντική στιγμή ήταν η στιγμή θέσης εφαρμογή της ε, ανταλλαγής πληροφοριών Schengen δεύτερης γενιάς. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα με νέες λειτουργίες, με νέα alerts, με νέες ειδοποιήσεις και έχει μεταφερθεί πλέον στο EULIS και έχει ε, πλέον καταστεί λειτουργικό. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην ε, Δυτική Αφρική, στην Κεντρική Αφρική και στην Ανατολική Αφρική έχει εφαρμοστεί ένα σύστημα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και είμαστε ευτυχείς που λειτουργεί σωστά το σύστημα αυτό. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές, για την έκθεση αυτή και για την συντομία σας, γιατί έχουμε πίεση χρονική. Και τώρα να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Ιτσιό. Ιτσιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώς. Και θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι με την έγκριση της νέας ε, των νέων κανόνων για το Σέγγεν λαμβάνει μεγαλύτερη ε, ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρακολούθηση του κεκτημένου και ελπίζω λοιπόν αυτό να βελτιώσει την κατάσταση. Κυρίως ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά σύνορα, περιορίστηκαν οι ροές χάρη στην επιχείρηση ασπίδα, χάρη σε αυτούς τους πολύ αυστηρούς ελέγχους. που δεν θα έχουν επιβαρυντική επίπτωση για αυτούς που πρέπει να έχουν διεθνή προστασία και κινούνται μέσω των μεταναστευτικών αυτών οδών. Η, Ευρωπα... η αστυνομία καλή να ελέγχει λοιπόν τα πάντα, όχι μόνο τους ε, μετανάστες, αλλά και το κατά πόσον τηρούνται οι σχετικές ε, νομοθεσίες. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση αυτή προασπίσει εκ νέου την προσάρτηση της ε, Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σέγγεν. Και ελπίζω να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ο κ. Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η τρίτη έκθεση που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάμαι ότι στην πρώτη έκθεση αναφέρθηκαν και περιληφθήσαν πολλά αρνητικά στοιχεία για την ε, Ελλάδα. Επί την σημείο εισόδου για πολλούς λαθρομεστάναστες, Δυστυχώς αυτό εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη σημερινή κατάσταση και κοιτώντας τι γίνεται στην Ελλάδα, επειδή είναι και καλοκαίρι, τα πράγματα κατά πάσα πιθανότητα στα θαλάσσια σύνορα θα είναι δύσκολα. Ρωτώ λοιπόν το εξή. Θυμάμαι ότι η πρώτη έκθεση συμπεριλάμβανε αρνητικά σχόλια, στη δεύτερη έκθεση είχαν βελτιωθεί πολύ τα σχόλια αυτά και η κατάσταση και τώρα στην τρίτη έκθεση αναφέρεται ότι είναι σταθερή η κατάσταση, ότι είναι λιγότερε οι συλλήψει. Και αναρωτιέμαι αν στην επόμενη έκθεση και σε αυτή την έκθεση θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια σχόλια θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των χωρών και ιδιαιτέρως τη συνεργασία της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση ή τοποθέτηση της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, κατά πόσον έχει βελτιωθεί και για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το χώρο Σέγγεν με καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Ζανόκα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέφερε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Είναι θετικό αυτό. Να εκφράσω και εγώ την ελπίδα ότι θα εισακούσει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να θέσω ερώτηση, αλλά να υπογραμμίσω ότι χαίρομαι που είναι πολύ θετική η έκθεση και νομίζω ότι είναι και θετικέ οι εξελίξεις και επιτυχής η εξέλιξη του Frontex. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τρίτη έκθεση αυτή. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μοζάμερ για να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Έντσιο, να σας πω ότι εμείς δηλώνουμε μείωση των ατόμων. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Αλλά ασφαλώς και θα πρέπει να δίδεται πρόσβαση στις διαδικασίες ατησής για ασυλό. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές. Δεν ε, υπογραμμίζεται, δεν διευκρινίζεται ωστόσο ρητά για το αίτημα του κυρίου Παπα-Νικολάου να αναπτύξουμε παραπάνω σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία. Πάντα είναι, ξέρετε, ευαίσθητο θέμα το πόσες πληροφορίες συμπεριλαμβάνουμε στην έκθεση, γιατί προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο κεκτημένο του Σέγγεν. Προφανώς χρειάζεται συνεργασία και με τρίτες και βλέπουμε, για παράδειγμα, το κεφάλαιο για τι θεωρήσει. Ε, και για την επανειστοχή. Προσπαθούμε όμως να περιοριστούμε στην αυστηρή εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά προφανώς και η συνεργασία με την Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την διασφάλιση των συνόρων. Ελπίζω να απάντησα έτσι στις ερωτήσεις που απευθυνθήκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο σημείο για την Επιτροπή Αγνοωμένων στην Κύπρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των αγνωμένων στην Κύπρο πάντα απασχολούσε ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΛΥΠΕ, όπως ε, προκύπτει και στα ψηφίσματα του 2007 και 2008 και το 2011 προσφάτως. Το Δεκέμβριο του περασμένου έτος, μία αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Αγγιλάρ επισκέφθηκε στην Κύπρο και είχε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Αγνοωμένων στην Κύπρο που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Αγνοωμένων στην Κύπρο είναι το κατεξοχήν ενδεγμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών που έχει διοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για να εξετάσει τους αγνοούμενους ε, ε, από το 2004 και μετά. Κατά τις επισκέψεις αυτές η αντιπροσωπεία της ΛΥΜΠΕ επιτόπου είδε την δουλειά και που έχει γίνει και θα ζητήσω από τα τρίτη μέλη να μιλήσουν από καθένας. Τους Αριστοτέλους from the Greek Cypriotic member and Mr. Paul Henry Hardy the third member appointed by the... Τα τρία μέλη θα μας ε, δώσουν μια παρουσίαση για το έργο της Επιτροπής Αγνωμένων και για τις μελλοντικές τους προοπτικές. has been announced by our colleague, Mr. Carlos Κύριος Σε ποιον θα δώσουμε τον λόγο καταρχήν. Είσαστε μάλλον που διόρισε ο ΙΕ. Κύριε Πολ Ανρή. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι με μεγάλη τιμή παρίσταμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο, στις Βρυξέλλες, για να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για την πρόοδο των εργασιών μας στην Κύπρο. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Θα ακούσω κάποια σημεία. Οι συναδελφοί μου θα συμπληρώσουν και σε λιγότερο από 15 λεπτά θα σας δώσω το λόγο για να κάνετε ερωτήσεις και να μπορέσουμε συνεχεία να τις απαντήσουμε. Όπως ξέρετε, από πιο σύγχρονες συγκρούσεις όπως την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Ιράκ, στη Συρία σήμερα, όταν χιλιάδες ε, παιδιά, γυναίκες, ε, γη, κόρη δεν έρχονται σπίτι για φαγητό, μετά τη σύγκρουση θα πρέπει να υπάρξει η διαδικασία ε, συμφιλίωσης γιατί αν οι αγαπημένοι σου λείπουν ε, για 10, 15, 20 χρόνια, αυτό το κενό που σου αφήνουν δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Οποιοςδήποτε έχει έναν αγνοούμενο στην οικογένεια, ο μόνος για να, τρόπος για να βρει ειρήνη είναι να βρει τη σωρό του αγαπημένου του και να την θάψει με τιμή. Ε, α, αλλιώς χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει συμφιλίωση, όπως παραδείγματος χάρη στη Βοσνία. Ε, η δουλειά που κάνουμε δεν είναι επιστημονική, δεν είναι τεχνική. Προσπαθούμε να δώσουμε στους Κύπριους την ευκαιρία να γιατρέψουν ένα από τα πιο βαθιά τραύματα της πρόσφατης ιστορίας τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Έχουμε τρία μέλη στην Επιτροπή μας, έναν Ελληνοκύπριο, έναν Τουρκοκύπριο και ένα τρίτο μέλος που διορίζει ο ΙΕ, έχει μια εντολή που του δίδεται που του δόθηκε από το 81 από τρία ψηφίσματα του, ε, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2006 ως το 2013 ξεκινήσαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για να ανακτήσουμε χάρη στην βοήθεια μαρτύρων των γεγονότων ένα πρόγραμμα ανάκτησης, εκταφής, εντοπισμού και επιστροφής της ορού. Υπάρχουν 2.000 ένα αγνοούμενη στην επίσημη λίστα που συμφώνησαν και οι δύο πλευρές. 978 έχουμε βρει από τους 2001, που είναι το 45% όλων των αγνοωμένων. Και από τα 2001 αγνοούμενα άτομα, έχουμε βρει και έχουμε επιστρέψει συνολικά στις οικογένειές τους 4.003 άτομα. 90 με 92% του προπολογισμού μας το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε αυτές τις επιτυχίες που σας ανέφερα. Ο βασικός μας δωρητής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δουλειά του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας και η υποστήριξη που μας δίνετε είναι πολύ σημαντικά για σας. Έχουμε λάβει 9,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια. Σήμερα έχουμε 6 επιστήμονες που δουλεύονται στα εργαστήριά μας που δουλεύουν στα εργαστηριά μας και επιτόπου έχουμε 19 άτομα, 7 ε, στο βορρά, 2 στο νότο, που εκτάφουν, 5 ε, Τις όλους πέντε άτομα βρήκαμε στη Λευκοσία πρόσφατα. Έχουμε μάθει πολλά σε ό,τι αφορά την ανάκτηση, την εκταφή, την ταυτοποίηση και αυτά που βρήκαμε εμείς μπορούν να χρησιμεύσουν και σε άλλες επιτροπές ανά τον κόσμο, σε αυτή που λειτουργεί στο Ιράκ, που έχει τους περισσότερους αγνοούμενους στον κόσμο. Είχαμε πέντε επιστήμονες που ήρθαν για 18 μέρες σε εμά να μάθουν από τις διαδικασίες μας, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη ξεκινώντας αυτή την τεράστια προσπάθεια στο Ιράκ. Ήταν οι ιατροδικαστές αυτοί οι επιστήμονες. Θέλουμε να δώσουμε με απόλυτη σιγουριά όσο γίνεται, 99,999% τα βεβαιότητα, ότι τα λείψανα που δίνουμε σε μια οικογένεια ανήκουν όντως σε αυτήν την οικογένεια. Κάνουμε λοιπόν αναλύσεις με αίμα και κόκαλα. Με αυτόν τον τρόπο ε, εντοπίζουμε γρηγορότερα, το είδαμε αυτό και στο Σαράγεβο, τους αγνοούμενους. Το πρόβλημα είναι ότι τα κόκαλα στην Κύπρο είναι των ατόμων αυτών είναι παλιά, είναι ανακατεμένα με τα κόκαλα πολλών ανθρώπων. Κάνουν πέντε αναλύσεις ανά ε, πτώμα. Είναι 300 ε, ευρώ κοστίζει ανά δείγμα η ανάλυση. Έχουμε ένα προϋπολογισμό ε, δύο ετών που το χρησιμοποίησαμε όλο μέσα σε δέκα μήνες όμως. Ε, αυτά είναι τα βασικά μου συμπεράσματα. Με το σημερινό βαθμό, ρυθμό έχουμε εντοπίσει και επιστρέψει ο 20% όλων των αγνώμενων στην ε, Κύπρο και με το σημερινό βαθμό θα χρειαστούμε ε, την υποστήριξή σας τα επόμενα χρόνια. Το 20% δεν αρκεί για να σταματήσουμε, δεν αρκεί για την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα ψηλότερο ποσοστό, 50-60% και επομένως θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε το σημερινό ρυθμό. Ολοκληρώνοντας, Θέλω να σας πω ότι οι σημερινές προκλήσεις που έχουμε από πέρυσι τέλο πάντων είναι πρώτον να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό δουλειάς με τους 19 επιτόπου, 25 ε, επιστήμονες στα εργαστηρία, εκατοντάδες δείγματα κοκάλων στέλνονται, οχτών στέλνονται στο Σαράγεβο για τακτοποίηση και έχουμε 80 με 100 τακτοποίησεις ανά έτος. Μέχρι τον Ιούνιο είχαμε 71 ταυτοποίησεις προσώπων. Είναι η δεύτερη καλύτερη χρονιά μέσα σε... και το πετύχαμε αυτό το ποσοστό μέσα σε 6 μήνες μόνο. Για να κρατήσουμε αυτό το ρυθμό και θέλουμε να το κρατήσουμε, βασιζόμαστε στους μάρτυρες και στους πληροφοριοδότε. Συγγνώμη, πληροφοριοδότες, οι οποίοι όμως επειδή είναι παλιά η σύγκρουση, ε... είναι από τη δεκαετία του 70, ε, αυτοί πεθαίνουν. Ε, ε, για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό μας. Ε, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει 2,2 με 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να το αυξήσουμε αυτό το ποσοστό κατά 300.000 ευρώ το χρόνο, που είναι 12% αν θέλουμε να κρατήσουμε το σημερινό ρυθμό, δεδομένου του ότι τα οστά είναι παλιά, είναι ανακατεμένα με τα οστά πολλών ανθρώπων, πολλών ανθρώπων ε, μεταξύ τους και πρέπει να κάνουμε πολλές ε, αναλύσεις από ό,τι είχαμε προκλέψει αρχικά. Τρίτη προτεραιότητα είναι η πολιτική να μείνει έξω από τη δουλειά μας. Είμαστε, βουλιάζουμε μέσα στην πολιτική, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε την πολιτική απ' έξω. Και μόνο με ένα... Και αυτός είναι ο μόνος μηχανισμός που δουλεύει στην Κύπρο σήμερα για αυτό το θέμα. Και Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η συνεισφορά σας, της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου σας είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τις οικογένειες αυτές, αλλά και για το μέλλον της Κύπρου. Είναι σημαντικό για την ειρήνη και την συμφιλίωση. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς να διεκπαιρεώσουμε αυτό το τεράστιο θέμα των ε, αγνοούμενων. Αν παραμείνουν αγνοούμενοι αυτοί, θα έχει τρομακτικές ε, πολιτικές συνέπειες για το μέλλον της Κύπρου αυτό. Η κυρία Γκυλτέν ε, Κιουτσούκ, αν θέλει να προσθέσει κάτι, παρακαλώ. Η κυρία Γκυλτέν Κιουτσούκ, που είναι Τουρκοκύπρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό. Θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεχίσετε να, υποχρε... να υποστηρίζετε το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να είναι βιώσιμο το έργο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο για την Κύπρο. Είναι το μοναδικό έργο που εμπλέκει και τις δύο κοινότητες που προσπαθεί από το 1963 να δώσει μια απάντηση στην αγωνία και στον πόνο των οικογενειών. Μισό αιώνα λοιπόν χρειάστηκε μέχρι ότου να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί ε, βάσει της πραγματικότητας που επικρατεί στην Κύπρο. Ξεκίνησε το 2006 και πιστεύω ότι όπου υπάρχει βούληση υπάρχει και τρόπος να ε, πετύχουμε τα αποτελέσματα. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει αποτελεσματικότητα χρειάζεται πολιτική υποστήριξη η οποία μας παρέχεται. Αλλά θα πρέπει να μην δοθεί και πολιτικός χαρακτήρας και αυτό ε, τηρείται είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι δύο κοινότητες, γιατί απευθύνεται και αντιμετωπίζει θέματα και των δύο κοινοτήτων. Επίσης, η Επιτροπή λειτουργεί με συνένεση και αυτό μας ε, επιτρέπει να λειτουργούμε και το έργο βασίζεται σε ε, μια διαδικασία απόρριτου και βασιζόμαστε σε ε, αυτόπτες μάρτυρες. Ψάχνω λοιπόν Ελληνοκύπριους και ο Ελληνοκύπριος ψάχνει τουρκοκύπριους αγνοούμενους. Άρα χρειάζεται συνεργασία και εμπιστοσύνη με βάση την καλή θέληση προκειμένου να πετύχουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μοντέλο που θα έχουμε δημιουργήσει και για τη μελλοντική Κύπρο. Όπως σας είπα, πρόκειται για ένα ευαίσθητο και πολυδιάστατο θέμα πολιτικά, έχει διάσταση, ανθρωπιστική διάσταση, ε, οικονομική διάσταση, διάσταση ανθρώπινου δυναμικού και πολλές άλλες. Το πιο, αν θέλετε, δύσκολο κομμάτι είναι αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση. Το έργο αυτό είναι ένα έργο το οποίο ζει και αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Προσαρμόζεται. Προσπαθούμε να το επιταχύνουμε, δε. Επειδή, όπως σας είπα, έχει περάσει και μισός αιώνας. Ο κόσμος, οι αυτόπτες μάρτυρες σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή, πεθαίνουν. Είναι μεγάλη πίεση από τις οικογένειες να επιταχύνουμε. Και γι' αυτό λοιπόν επανασχεδιάζουμε το πρόγραμμα αυτό. Με τον τρόπο αυτό ανακύπτουν επιπλέον οικονομικές ανάγκες. Χρειαζόμαστε υποστήριξη. Το σχέδιο λοιπόν έχει και βάσει σε τέσσερις φάσεις. Εκταφή, ανθρωπολογική, ταυτοποίηση και επιστροφή λειψάνων. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή των λειψάνων, να σας πω ότι είναι το πιο συναισθηματικό κομμάτι, γιατί στην περίπτωση αυτή για πρώτη φορά οι οικογένειες βλέπουν τους αγαπημένους τους υπομορφή οστών. Η διάσταση που λείπει είναι η δίωξη, αν θέλετε. Έχει μπει και αυτή σιγά σιγά στο πλαίσιο. Όπως σας είπα, το σχέδιο αυτό ζει και αναπτύσσεται και στην εξέλιξή του προσπαθεί να προσαρμοστεί βάσει και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των σχετικών αποφάσεων το δικαστήριο ζητά και από τους εισαγγελείς και από την αστυνομία να κάνουν σχετικές ερευνές. Είναι σημαντικό και το σκέλος αυτό. Έχει στεφθεί με επιτυχία το, το πρόγραμμά μας. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχει περάσει και μισός αιώνας. Είναι πολύ καλή η ταχύτητά μας, η αποτελεσματικότητά μας και με χαρά σας ανακοινώνω ότι η χρηματοδότησή σας ε, πιάνει τόπο. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για την υποστήριξή σα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρο και τώρα τρίτος ε, ομιλητής, ο κύριος Άριστος Αριστοτέλους από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κάλυψαν τα περισσότερα, αλλά πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε μπορέσαμε σήμερα να έρθουμε εδώ, να εμφανιστούμε ενώπιον τη Επιτροπή σα. Βεβαίω και εκτιμούμε πάρα πολύ το ενδιαφέρον σα, αλλά και τη βοήθειά σα όσον αφορά την ε, όλη αυτή η υπόθεση αυτή τη ανθρωπιστική αποστολή. Οπωσδήποτε. Σε εμά προβλέπουν οι Κύπροι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ και στους άλλους διεθνείς φορείς, διεθνείς φορείς οι οποίοι για την υπόθεση αυτή. Επίσης, μπορώ να σας αναφέρω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα με που έχω ασχοληθεί, τα οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τη συνέχιση των δικοινοτήτων, την, βοηθήσουν την υπόθεση ειρήνης στην ε, Νήσο. Επίσης, από πλευρά επιστημονική να σας πω, αλλά να σας πω επίσης και ποιε είναι για το μέλλον, τι αποτέλεσμα έχουμε αποσπάσει μέχρι σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την πτυχή ειρήνευση, έτσι όπως προχωρούμε, συνεργάζονται οι δύο κοινότητες. Έχουμε επιστήμονε και από τις δύο κοινότητε που συνεργάζονται. Και Πρόκειται για μια προσπάθεια την οποία εκτιμούν ιδιαίτερως οι πολιτικοί και από τις δύο πλευρές. Επίσης έτσι αποτελούμε ένα παράδειγμα προς ε, μίμηση αλλού στον κόσμο όπου επίσης υπάρχουν σύγκρουσεις. Δεν είναι τυχαίο το ότι αναφέρθηκε ε, στην ε, υπόθεσή μας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και το ανέφερε λέγοντα ότι αποτελεί παράδειγμα προ μίμηση. Ούτε επίση είναι τυχαίο ότι από άλλε περιοχέ όπου σοβούν σύγκρουσει έρχεται ο κόσμο ή στην Κύπρο να παρακολουθήσει τι γίνεται και πώ ω Επιτροπή ε, έχουμε στη συνεργασία που σα είπα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ε, φέρουμε πέρα σε αυτό το ανθρωπιστικό έργο. Τώρα, όσον αφορά την επιστημονική πτυχή του εγχειρήματό μα, οφείλω να σα πω ότι Πέραν των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από πλευρά επιστημονική προσέγγιση, επίσης έχουν έτσι ανοίξει καινούργιε λεωφόροι όσον αφορά την επιστήμη της εκταφής, όσον αφορά την αρχαιολογία και την ανθρωπολογία. Και γι' αυτό και πολλοί διεθνεί φορεί έχουν απευθυνθεί ει του ε, επιστήμονε με του συνεργαζόμαστε και του ζητούν να υπάρξει συμβολή στις ξενόγιες προσπάθειε που γίνονται. Δεν είναι εύκολο αυτό το έργο. Αλλά κατά τη γνώμη μας θα πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα αφορά τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματο, προλαλήσαντες σας είπαν. Πάνω κάτω τι ισχύει, πάντω λόγω τη καινούργια δομή που πρόσφατα υιοθετήσαμε, τώρα είμαι η θέση να αποσπάσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και όσο περισσότερη ταυτοποίηση έχουμε, τόσο περισσότερες οικογένειε θα ανακουφιστούν. Έτσι θα μπει ένα τέρμα στο βάσανό τους, στον πόνο, στην οδύνη που αισθάνονται αισθανόνται για τόσο καιρό. Οπότε ο σκοπός μας είναι ακριβώς αυτό, το να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό των εργασιών μας. Θα είπα τώρα τι δυνατότητες έχουμε για να πάμε σε περισσότερες ταυτοποίησεις και έτσι να έχουμε την επιστροφή των σωρών στις οικογένειες. Ακόμα βέβαια έχουμε δουλειά μπροστά μας. Βεβαίως είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πάντα μπορεί, επειδή έχετε βελτίωση συνεργασία και πάντοτε ε, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερους πόρους. Βέβαια, υπό την συγκυρία της κρίσης, δεν είναι τόσο εύκολο έτσι να βοηθήσουμε. Και πρόκειται επομένω για πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε το οικονομικό και επίση ελπίζουμε ότι με τη βοήθεια διεθνών φορέων όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάρα πολύ σημαντικός βοηθός μας, θα φέρουμε εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Και βέβαια υπολογίζουμε και στην βοήθεια της δικής σας επιτροπής που επανειλημμένα αποδείξατε ότι μπορεί να βοηθήσετε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Έτσι θα βοηθεί ακόμη περισσότερο η υπόθεση η ειρήνη, έτσι θα ελαφρύνουμε περισσότερο την οδύνη αυτών των ανθρώπων. είναι το ανθρωπιστικό το έργο μας, αλλά βεβαίως και υπάρχει και η πολιτική πτυχή την οποία συζητήσαμε στην αρχή. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Okay. Now, heard... Πρόεδρος. Τόσο μικροφόνο. Και τώρα ήρθε η ώρα να λάβουμε το λόγο τα μέλη της Επιτροπής μας για παρατηρήσεις. Κύριε Τρενταφυλλίδης, ο πρώτος. Much καλωσορίζω τα τρία μέλη της Επιτροπής και τα ευχαριστώ για τα θαυμάσια αποτελέσματα που πέτυχαν και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ τους για αυτό το τόσο κλεπτό θέμα. Όταν επισκεφτήκαμε την Κύπρο το Δεκέμβριο ως Επιτροπή ΠΥΜΠΕ, τότε μόνο συνειδητοποίησαμε τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει στα πλαίσια αυτού του προγράμματος σε όλα τα επίπεδα, συνεργασία, μη πολιτική, σε όλα τα επίπεδα κτλ. Και για να γίνει αυτή η δουλειά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται μια απαραίτητη πόρη. Επομένως, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι ως Επιτροπή καλό θα ήταν να υποβάλουμε ένα αίτημα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να αναδιανέμει κάποια από τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται και που υπάρχουν για την τουρκο-κυπριακή κοινότητα, για να δοθούν σε αυτήν την Επιτροπή. Σας ζητώ λοιπόν να κάνετε επίσημη αίτηση στην Επιτροπή Προπολογισμών, τόσο ώστε αυτά τα 300, οι 300.000 ε, ευρώ επιπλέον που χρειάζονται ανά έτος να βρεθούν ούτως ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το συντομότερο δυνατόν, γιατί καταλαβαίνω ότι θα χρειαστούν χρόνια, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Ελπίζω να σημειώσατε την πρότασή μου, Πρόεδρε. Και αν χρειάζεται η συνένεση Επιτροπής μας, θέσετε αυτό το ερώτημα στην ε, Επιτροπή, στα μέλη της Επιτροπής, ώστε να το υποστηρίξουμε. Και να το ψηφίσουμε βέβαια. Εντάξει, το σημείωσα κυρία Τρενταφυλλίδη. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ε, που έγινε πέρσι και για μια ακόμη φορά θεωρώ ότι ε, είναι ανθρωπιστικό το δράμα των αγνωμένων και συγχαίρω την Επιτροπή, την Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων γιατί κάνει μια αξιόλογη δουλειά και μάλιστα στέλνει και ένα μήνυμα συνεργασίας με την ε, συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να χτίσουμε μαζί ε, ένα κοινό μέλλον. Ε, εκείνο το οποίο πραγματικά με έχει απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ το θέμα των αγνωμένων είναι η δυστοκία που παρουσιάζεται όταν υπάρχει ακριβώς προσπάθεια για να γίνει η διερεύνηση σε στρατιωτικές περιοχές. Και αυτό προέκυψε και στην συνάντηση που είχαμε με την Ηνωμένα Έθνη και με άλλους αρμοδίους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Τέθηκε επιτάπητος το θέμα ότι υπάρχουν στρατιωτικές ζώνες και δεν ρωτούμε υπάρχει ένας οδικός χάρτης και έχει γίνει ένας χάρτης όπου να φαίνεται σε ποιες περιοχές πιθανόν να υπάρχουν ακόμα σωρία γνωμένων ή σκελετοί και τέτοια για να μπορεί να διερευνηθούν συγκεκριμένα σημεία για να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι σε αυτή την περιοχή δεν μπορεί να πάει ιδέα γιατί είναι στερεωτική περιοχή. Μας έχει καταγγελθεί ότι υπάρχει μια διαρκής μετατόπιση και καθορίζονται νέες στρατιωτικές ζώνες. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο στην προσπάθεια της Επιτροπής. Θα ήθελα να δω από τώρα και στο εξή τι γίνεται για αντιμετώπιση αυτού του καυτού προβλήματος και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Το δεύτερο αφορά την Τουρκία. Παρακολούθησα εδώ και πολλά χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης το θέμα των αγνωμένων. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να δώσει στοιχεία και δυστυχώς υπάρχει μια προθυμία ε, για να δώσει αυτά τα στοιχεία. Και ε, πολλές φορές ε, πρέπει να γίνει έρευνα και στην ίδια την Τουρκία, τη χώρα της Τουρκίας. Και εδώ υπάρχει μια προθυμία. Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, να διαβεβαιώσω ότι από δικής μας πλευράς ε, θέλουμε πραγματικά να διερευνηθεί το, η τύχη του κάθε αγνώμενου, γιατί αυτό είναι δικαίωμα των οικογενειών και παρόμοιε εκθέσει έχουν γίνει για πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη, στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αναφέρει το δικαίωμα να μάθουν τι απέγινα. Μια απασχολία όμως και μια άλλη πτυχή που είναι πέραν από το mandate του όρου εντολή τη ΔΕΑ. Πρόσφατα δημοσιεύματα σε κυπριακέ εφημερίδε έχουν δείξει ότι σε πάρα πολλούς σκελετούς και σε πάρα πολλά κεφάλια που έχουν εντοπιστεί και υπήρχαν φωτογραφίε στον τύπο, πραγματικά φαίνεται ε, ότι αυτά τα άτομα που χάθηκαν έχουν υποστεί βασανιστήρια και ε, με έχουν πλησιάσει συγγενείς αγνωμένων και διαμαρτυρήθηκαν γιατί στα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις περιπτώσεις που έχουν διακριβωθεί οι τύχες τους καταγράφεται θάνατος από άγνωστα αίτια και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι άδικο γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χάθηκαν διασκεδάζοντας δεν χάθηκαν πηγαίνοντα σε μια εκδρομή. Χάθηκαν σε έναν πόλεμο που έγινε το 1974, σε μια εισβολή. Και διερωτούμε ρωτούμε αυτά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τους Τουρκοκύπριους και για τους Ελληνοκύπριους γράφουν ακριβώς σαν αιτία θανάτου άγνωστη αιτία. Θα ήθελα να ξέρω αυτά τα πιστοποιητικά πώς εκδίδονται και αν είναι δυνατόν να μας παρουσιαστούν. Κύριε Πρόεδρε, ε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδότηση και τη στήριξη που παρέχει στη ΔΕΑ. Νομίζω ότι γίνεται μια δουλειά η οποία τιμά τους Κύπριους τολμώ να πω με ένα συμβολισμό που έχει μια παγκόσμια σημασία. Σπάνια κατάφεραν ε, μετά από συγκρούσεις ε, λαοί, κοινότητες να συνεργαστούν τόσο άψογα στο να βρεθούν τα λείψανα των νεκρών ε, ενός πολέμου. Ε, θέλω ιδιαίτερα να, να συγχαρώ το τρίτο μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής, τον κύριο Ανρή, που προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι ως Κύπριος σε αυτή τη δουλειά. Θα θυμίσω και τον προηγούμενο τρίτο μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Ζηρότο, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια πρόσφερε πολύ μεγάλες υπηρεσίες ε, σε αυτή τη διαδικασία και στην Κύπρο. Ασφαλώς την κυρία Κουτσούκ εκ μέρους της τουρκοκυπριακής κοινότητας και τον φίλο μου τον Άριστο, τον Αριστοτέλους, για την δουλειά που κάνει. Εγώ θέλω να προσθέσω την εξή πτυχή Νομίζω ότι αυτή η δουλειά που γίνεται πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διαχυθεί μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Νομίζω ότι είναι λίγο απομονωμένη η δουλειά που γίνεται ε, μέσα στα εργαστήρια. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τρόπους να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις κοινότητες αυτή η δουλειά που επαναλαμβάνω έχει τον παγκόσμιο συμβολισμό που έβαλα να μπορεί να περάσει στον κόσμο ε, για να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει πέραν της ανέβρεσης των οστών των αγνοωμένων που είναι η, δυνατότητα των κοινοτήτων όπως άψογα συνεργάζονται σε αυτή τη δουλειά να μπορέσουν και στο μέλλον με μια λύση στο Κυπριακό να ζήσουν μαζί αφού κατανοήσουν πρώτα απ' όλα την, ότι ο πόνος δεν, δεν, έχει, δεν έχει καταγωγή. Ε, το τελευταίο που έχω να πω Νομίζω ότι είναι καλό ο τουρκικός στρατός, θα πάω σε μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή, δεν μπορεί παρά να, έχει στα, στα αρχεία του ε, πληροφορίες για το πού έχουν ταφεί ε, νεκροί του πολέμου. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολλά. Ενώ τώρα αυτή η δουλειά γίνεται ε, από απλούς πολίτες τους οποίους κανείς πρέπει να συγχαρεί και κατηδίαν και δημόσια κάποτε και με κίνδυνο της ζωής τους να βρουν πληροφορίες και να τις δώσουν στη ΔΕΑ ενώ θα, θα έρχονταν μια μαζική πληροφόρηση αν άνοιγαν τα, τα αρχεία του, του στρατού της Τουρκίας. Με αυτά εγώ κλείνω ξανά συγχαίροντας και ευχαριστώντας και τα τρία μέλη για την ε, πολύ μεγάλη και χρήσιμη δουλειά που κάνω. Ευχαριστώ. Mr. Bronx. Thank um, Ο κ. Μπρόγκς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσοι και τι ποσοστό των αγνοωμένων και λειψάνων προέρχονται από τις δύο κοινότητες. Κατά δεύτερον υπάρχουν ενδείξεις για το κατά πόσον ή πόσοι εξ αυτών ε, έχουν ε, δολοφονηθεί από στρατιώτες ή από αντάρτες, από άτομα που δεν ανήκαν στις στρατιωτικές δυνάμεις και επίσης ε, έχετε βρει τα κριτήρια για, με τα οποία επιλέχθησαν τα θύματα, ποιοι ήταν, μπορούν να γίνουν κάποιες γενικές διαπιστώσεις για τα θύματα και θα υπάρξει μια έκθεση η οποία θα ε, γίνει στην, όταν τελειώσει η διαδικασία αυτή, όχι σύντομα δηλαδή, και ένα ρητορικό ερώτημα να θέσω θα μπορέσει να υπάρξει πραγματικά ε, να κλείσει το θέμα αυτό, ακόμα και όταν βρίσκονται τα λείψανα, όταν ε, δεν θα μπορέσουν να θάψουν στα λείψανα τους ε, στο βορρά της Κύπρου. Και τι δυνατότητες υπάρχουν να συζητηθεί αυτό με την Τουρκία και όχι με τους Τουρκοκύπριους. Μίλησα με κάποιους εξ αυτών και πολλοί εξ αυτών είναι κατά τη κατοχή και νομίζω ότι το γεγονό ότι εκπροσωπούνται και οι δύο κοινότητε στην Επιτροπή αυτή είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Τι συνεργασία έδωσαν οι τουρκικέ αρχές ε, στο Βορρά και από την τουρκική κυβέρνηση. Έχω κάποιες ενδείξεις φυσικά από άλλα μέλη. Ευχαριστώ. Ο κ. Σοφοκλέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, τρία σύντομα σχόλια και μία ερώτηση. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι συμφωνούμε όλοι ότι έχετε ένα δύσκολο έργο να επιτελέσετε σαν Επιτροπή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τούτο. Το δεύτερο μου σχόλιο είναι ότι επίσης όλοι συμφωνούμε ότι ίσως είναι η τραγικότερη πτυχή μετά από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στο θέμα των αγνωμένων. Όσα χρόνια και να περάσουν, αν δεν υπάρξει η διακρύβωση της τύχης των αγνωμένων και Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να κλείσει. Το τρίτο μου σχόλιο είναι μία κριτική προς την Επιτροπή. Θετική όμως κριτική. Δηλαδή έχουμε μία Επιτροπή η οποία έχει την έξωθε εξαιρετική καλή μαρτυρία. Και μιλώ για τη συγκρότησή της. Εκπροσωπείται από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών στην ουσία και από τις δύο κοινότητες. Και το θεωρώ σημαντικό πολιτικό εχείρημα και επίτευγμα. Η ερώτηση όμως, όμως είναι η εξής παρότι δεν θα ήθελα πραγματικά σαν Ελληνοκύπριος Ευρωβουλευτής να πολιτικοποιήσω, όπως είπατε, το ζήτημα που χρειάζεται πολλές φορές. Η Τουρκία σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλεται συνεργάζεται μαζί σας. Δηλώσεις που κατά καιρού έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν ανακοινωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα αναγνωμένο. Ή αυτό που έχει λεχθεί από συνάδελφο μου ότι Υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές, στρατιωτικές περιοχές που δεν δίδεται η δυνατότητα, ευκαιρία να κάνετε την δουλειά σας καλά. Πώς αξιολογείτε αυτή την θέση της Τουρκίας και βέβαια, κλείνοντας σε επιμέρους σημαντικό ερώτημα, που επίσης έχει λεχθεί και μας έχει και με έχει απασχολήσει, πόσοι έχουν δολοφονηθεί μέσα από την διερεύνηση, όχι πόσοι έχουν σκοτωθεί μέσα από τη διερεύνηση και την εξακρίβωση, τον στοιχείο και ότι άλλο σκοτώνεται κανένα σε μια μάχη που δεν πρέπει να γίνεται και άλλον δολοφονείται βάναυσα και απάνθρωπα που είναι ό,τι χειρότερο. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και επειδή έχει προχωρήσει και η ώρα, θα είμαι σύντομη, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις Ήμουν και εγώ μέλος της ε, αντιπροσωπείας πέρσι. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό πώς υπό τόσο δύσκολες συνθήκες κάνετε τη δουλειά σας και νομίζω ότι όλοι ήταν πολύ εντυπωσιασμένοι. Όλα τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας είμαι βέβαιη ότι όλοι θα ταχθούν υπέρ της συνέχισης του έργου σας. Ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι η πρόταση τρινταφυλλίδη είναι πάρα πολύ πετυχημένη να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια τα οποία δεν αξιοποιούνται στην παρούσα φάση, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια πραγματική συμβολή στην ειρήνευση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και δεν καταλαβαίνω την στάση της τουρκική πλευράς να μην ανοίξει τα αρχεία της, να μην δώσει πρόσβαση στις στρατιωτικά κατεχόμενες ζώνες, γιατί με τον τρόπο αυτό αποτρέπουν και το να μάθουν και οι Τουρκοκύπροι κάτι για τους ε, συγγενείς τους και Ακούσαμε ακριβώς από τους τουρκοκύπριους την ε, αποστολή ότι είναι δυσαρεστημένοι. Και υποθέτουν ότι στις στρατιωτικές κατεχόμενες ζώνες είναι πάρα, πολλές, πάρα πολλά τα λείψανα ακόμα. Και ναι, ο τουρκικός θα πρέπει να ανοίξει τα αρχεία του και θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε από την Επιτροπή μας για τη συνέχεια της χρηματοδότησης της Επιτροπής σας. Ελπίζω να υπερψηφίσουμε ένα σχετικό ψήφισμα. Πρόκειται για ένα ειρηνικό έργο, σχέδιο. Και ακούτε και από τα άτομα που πήραν το λόγο εδώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνει εκτός πολιτικού χαρακτήρα το θέμα αυτό γιατί η τουρκική πλευρά σε αυτή τη ε, φάση θα αντιδράσει υπερευαίσθητα αν ασκηθεί οποιαδήποτε κριτική, η οποία πιστεύω παρόλα αυτά ότι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Okay. Μάλιστα. Ακούστηκαν διάφορες ερωτήσεις. Ακούσαμε το, την πρόταση του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Δεν ακούμε για πρώτη φορά τη σημασία που δίνεται στο ότι τα ποσά που θα πρέπει να αποφασιστούν με βάση τις δημοσιονομικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος. ένα πρόγραμμα που έχει υποστήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει όσους έχασαν και να ζητούν τους αγαπημένους τους. Τη στιγμή της διαίρεση τη της Κύπρου. Ψάχνουν λοιπόν τους αγνοούμενους. Καταγράφουμε λοιπόν την πρόταση και νομίζω ότι είναι και η ώρα να ακούσουμε την απάντηση των ομιλητών μας. Θέλετε να απαντήσετε στα όσα ακούσατε. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε κι εσείς με τη σειρά σας, γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος. Αμέσως μετά έχω μια συνάντηση με την επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία ούτως ή άλλως, άρα δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν κυρίε και κύριοι. Όλες οι ερωτήσει σας δείχνουν ότι ξέρετε πολλά για το θέμα. Υπάρχουν τέσσερις τομείς τη σα. Η πρόσβαση στις στρατιωτικέ περιοχές του Βορρά, ε, συνθήκες θανάτου, δεύτερον, βασανίστηκαν, δεν βασανίστηκαν, τι αποδεικτικά στοιχεία έχουμε. Τρίτον, η δουλειά αυτή να βγει από τα εργαστήρια, να γνωστοποιηθεί να τη μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι τρεις τομείς. Και το ερώτημα που ακούστηκε για τα ποσοστά των αγνοούμενων ανακοινότητα. Αυτό συνδέεται και με τις συνθήκες θανάτου. Να σας δώσω αυτά τα λίγα νούμερα που έχουμε σήμερα. Έχουμε επιστρέψει 338 Ελληνοκύπριους από έναν αρχικό αριθμό 1590, 32-33%. Βρήκαμε επίσης 17 Τουρκοκύπριους από τους 502. Είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Υπάρχει μια δυσαναλογία δηλαδή. Βρίσκουμε περισσότερους Ελληνοκύπριους στο ΟΡΑ από ότι Τουρκοκύπριους στο Νότο. Και αυτή είναι μια από τις ανησυχίες μου. Να κρατήσω ε, περίπου τα νούμερα ισοσκελισμένα και ανάλογα με το συνολικό πληθυσμό. Αυτή η ισορροπία είναι σημαντική ούτως ώστε ε, η κυρία Κιουτσούκ να συνεχίσει να έχει την υποστήριξη ε, των τουρκοκυπριακών αρχών αλλά και του τουρκικού Υπουργείου. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Συνθήκες θανάτου. Δεν έχουμε εντολή να αναλύσουμε και να δώσουμε πιστοποιητικά για τις συνθήκες θανάτου. Όπως ξέρετε, στην Κύπρο. Υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Και οι δύο εισαγγελεί του Βορρά και του Νότου έχουν γραπτό συμφωνήσει ότι οι μάρτυρες θα έρχονται με πληροφορίε και δεν θα διώκονται. Εμείς θα έρχονται σε εμά. Και εμείς ε, θέλουμε να εντοπίσουμε και να επιστρέψουμε τα λείψανα, όχι να δούμε τις συνθήκε του θανάτου. Κρατάμε όλα τα αντικείμενα και τι σφαίρε και οποτεδήποτε τεθούν ρωτήσει στα πλαίσια της διαδικασίας του Στρασβούργου, θα απαντήσουμε με βάση τα όσα ξέρουμε. Αλλά δεν κάνουμε ανάλυση στο εργαστήριο, ε, στη σήμανση δηλαδή, για να δούμε αν κάποιος ε, πυροβολήθηκε ε, εκ του Η πρόσβαση σε στρατιωτικές περιοχές. Πολύ ξεκάθαρα πρέπει να απαντήσω από το 2006 ζητήθηκε πρόσβαση σε συγκεκριμένες στρατιωτικές περιοχές στο Βόρα. Το ζητήσαμε 22 φορές. Δόθηκε πρόσβαση και τις 22 φορές. Καμία άρνηση μέχρι στιγμής δεν είχαμε. Πάμε βήμα-βήμα, γιατί ο στόχος μας είναι η πρόσβαση. Δεν είναι η αντιπαράθεση ή το να προσκρούσουμε σε άρνηση. Τον Ιανουάριο φέτος ζητήσαμε για πρώτη φορά πρόσβαση σε ένα στρατόπεδο στρατιωτικό με σειρματόπλεγμα. Μας δόθηκε, είδαμε πέντε λείψανα. Ε, τον περασμένο μήνα δουλέψαμε ε, και εξήμαν των θυρών οι τρεις μας για να συζητήσουμε τα περαιτέρω βήματα για τις ιδιωτικές περιοχές. Και εμείς συμφωνήσαμε και εκείνοι συμφώνησαν ότι θα δούμε Αυτά είναι τα συγκεκριμένα μέρη που θα να ζητήσουμε πρόσβαση, με την τάδε σειρά κτλ. Συμφώνησαν δηλαδή και μεταξύ του. Έτσι λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία θα συνεχίσουμε. Διάδοση των στοιχείων που έχουμε, το συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε ισχύσει παρατηρήσει με τις δικέ σα. Θα θέλαμε να συζητήσουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία έκθεση που θα παρουσιαστεί και, στην Κύπρο αλλά και εδώ στη Βρυξέλλες, στην πλάση του Λουξεμβού. Αλλά είμαστε σε αρχικά στάδια αυτών των συζητήσεων για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικό και σε μια ε, δεύτερη φάση να το παρουσιάσουμε και σε σχολεία στην Κύπρο, στην Κύπρο ούτως ώστε η δουλειά αυτή να γίνει γνωστή και να, καταλάβει, να καταλάβουν και οι κοινότητες πόσο σημαντική και πόσο βαθιά είναι αυτή η δουλειά και πόσο σημαντική είναι και για τις δύο κοινότητες, ε, είτε είσαι Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος και πόσο μεγάλο το δράμα είτε είσαι Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος. Σας ευχαριστώ. Έχουν απαντηθεί πιο πολλά ερωτήματα. Θα κάνω μόνο κάποια σχόλια. Έγινε μια ερώτηση για την εκπροσώπηση της τουρκικής πλευράς. Εγώ είμαι ζώσα απόδειξη, γιατί εκπροσωπώ τους ε, τουρκοκύπριους και την τουρκική πλευρά. Είναι μεγάλη εκπροσώπηση. Το σχέδιο αυτό είναι δικοινωτικό. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη θέληση και της τουρκικής πλευράς. Υπάρχει λοιπόν υποστήριξη πλήρης υποστήριξη από πλευράς μου προς το project αυτό. Έγινε ένα σχόλιο για τα πιστοποιητικά θανάτου. Το θέμα της, ε, το, της αναλογικότητας, τα ποσοστά, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους αγνοούμενους. Οι Τουρκοκύπροι είναι όλοι άμαχοι. 28% γυναίκες και παιδιά, Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι, είναι όλοι 55% είναι στρατιωτικοί και περίπου 20 γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα, τελευταίο σημείο τώρα, ο κύριος Αριστοτέλους. Έχει το λόγο. Νομίζω ότι πολλά καλύφθησαν ήδη. διαρωτικά θα πρέπει να το δούμε, μακρόπνο το θέμα. Ακριβώ όπως το είπαν και οι περισσότεροι από του ε, ομιλητέ που ζητούν τον λόγο στον πρώτη χρηματοδότηση τέλο πάντων του εγχειρήματο, γιατί ε, είπαμε ότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να είναι ένα πράγμα προ μίμηση. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σαφέ σε όλου το πόσο δύσκολη αυτή η υπόθεση με το οποίο ασχολούμεθα, ε, γιατί ακριβώ οι στρατιωτικέ ε, περιοχέ ήταν ένα ζήτημα πάρα πολύ επίμαχο. Και μόνο κοιτάμε μπροστά ω Επιτροπή. Και ο συνέδελφος ο κ. σα σας είπε ότι συμφωνούμε στο ποιες περιοχές θα θεωρηθούν στρατιωτικέ και έτσι θα προχωρήσουν. Και αναλογιστούμε και τη σχετική άδεια για να δοθεί έγκριση να πάμε εκεί που θέλουμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Μια ναι, που έλαβα τελευταία στο λόγο, σας επαναλαμβάνω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την ανθρωπιστική προσπάθεια που έχει και αυτόν τον ειρηνευτικό χαρακτήρα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ όλους και εγώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Χατζηγεωργίου, έχει το λόγο ρώτησα εάν ο τουρκικό στρατό μπορεί να ανοίξει τα αρχεία του. Δηλαδή να μας πει ο ίδιο ο στρατός εάν ξέρει που υπάρχουν νεκροί. Εγώ λέω και η Εθνική Φρουρά εάν υπάρχει αυτό το αίτημα. Δηλαδή αυτό θα δώσει γνώση που είναι οι, οι, νεκροί του πολέμου. Any, any answer? Θέλει κάποιος να απαντήσει κύριε Αρνή. Όπως προανέφερα, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο με στρατηγικές περιοχές, όπου ως, περιοχή, Επιτροπή έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχουν κάποια υπολείμματα. Λείψανα. Οπότε εκεί επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας. Τώρα όσον αφορά τα αρχεία του στρατού, όντως και στο Στασβούργο έχει τεθεί αυτό το θέμα πολλές φορές δεν έχουμε κάνει τέτοια κίνηση ακόμη σε Επιτροπή. Διότι επικεντρώνουμε την προσοχή μας και τους πόρους μας και ανθρώπινους πόρους όχι στα αρχεία αλλά στους τάφους. Ασχολούμαι 23 χρόνια με αυτό το θέμα και στα Βαλκάνια επίσης ε, ήμουνα επικεφαλής στην αντίστοιχη υπηρεσία και για, τα αρχεία της K4 επίσης έχω ασχοληθεί. 18 χώρες ε, έστειλαν δυνάμεις ε, για την ΚΕΙΦΟΡ του, του Κόσοβου, του Κωσυφοπεδίου τέλο πάντων. Οπότε τελικά ανοίξαν τα αρχεία εκεί πέρα και ήταν όλε οι δυτικέ χώρες εκτό από τη Ρωσία. Και αφού κάναμε τρία, διαδήματα, μας, ε, μόνο τρεις χώρες. Μόνο τρεις χώρες μας έδωσαν κάποια στοιχεία. Μόνο τρεις χώρες. Υπόλοιποι... Και κανένα στρατός δεν θέλει να ανοίξει τέτοια αρχεία ούτε το ΝΑΤΟ βέβαια. Επομένω, Πολύ προσπάθεια, πολύ κακό για το τίποτα. Οπότε και γι' αυτό επικεντρώνουμε προσοχή μα σε αυτά τα, τα, σημεία, σε αυτού του τάφου. Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ, λέει ο πρόεδρο, αλλά πιέζει ο χρόνο. Και έχω τώρα και ένα ραντεβού με εκπροσώπου τη Λιθουανική Προεδρία. Αλλά και οι διερμηνεί πρέπει να αποχωρήσουν δούλεψαν μέχρι 6.30 έπρεπε να δουλέψουν και μας χάρισαν και κάποια λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.